Um, dear friends, dear friends, dear colleagues. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. Εξοχότητες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με την συνεδρίαση αυτή ξεκινάει η ένατη έκδοση ενός από του πιο σημαντικού ετησίου γεγονότος που λαμβάνει η χώρα στην Ευρώπη και που είναι οι Open Days, ανοιχτές μέρες, μέρες ελεύθερης προσέλευσης, όπου συμμετέχουν όλοι όσοι ασχολούνται με τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνάντηση μαζί και ότι η συζήτησή μας αυτή θα εμπλουτίσει το περιεχόμενο της πολιτικής μας συνοχής και θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και σε άλλες δράσεις. Θέλω λοιπόν εδώ εγκάρδια να υποδεχτώ εδώ και να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Γιέση Μπούζεκ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, εκ μέρους της Πολωνικής Προεδρίας την Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, την κυρία Ελισβιέντα Μπιενκόφσκα, που εξελέγει χτες στην Πολωνική Γερουσία, την κυρία Μπρέσο, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών και τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό βέβαια, τον Γιωχάνης Χάν, Επίτροπο για την Περιφερειακή μας Πολιτική. Αγαπητοί φίλοι, κάθε χρόνο μέσω των ημερίδων αυτών η Ευρώπη δίνει μεγάλη σημασία στην διάστασή της στην περιφερειακή και την τοπική ο ευρωπαϊκός δυναμισμός δεν μπορεί παρά να προέλθει από τις περιφέρειες, τις πόλεις και τους δήμους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτήν την καλή ε, περιφερειακή διακυβέρνηση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με την, την ε, κοινωνία των πολιτών. Κάθε χρόνο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί επιλέγουμε τα θέματα που θα συζητήσουμε. Και δεν μας εκπλήσει βέβαια το γεγονός ότι είμαστε εδώ σήμερα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί, για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη την οποία χρειαζόμαστε τόσο πολύ εμείς οι Ευρωπαίοι. Ε, προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους τρόπους, τα καλύτερα μέσα για να πετύχουμε και να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή μας έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε ε, ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια ανάπτυξη η οποία θα μας πάει πολύ πιο πέρα από εκεί που βρισκόμασταν πριν από την κρίση. Θέλουμε μια ανάπτυξη η οποία να μας βοηθήσει να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και την ανταγωνιστικότητά μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν βιώσιμη ανάπτυξη και για να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη πρέπει να είναι ευφύης, πρέπει να είναι βιώσιμη και πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλους. Και το χρειαζόμαστε όταν το νομοθετικό πακέτο για την περίοδο 2014-2020 της ε, πολιτικής συνοχής έχει έρθει στο τραπέζι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προβληματιστούμε πάνω σε αυτήν και να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτήν. Πριν από δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία που πιστεύω ότι θα το πετύχουμε γρήγορα. Με καλές σχέσεις με την Επιτροπή των Περιφερειών επίσης θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως θέλουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, συναποφασίζει με το Συμβούλιο για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τη νέα περίοδο πολιτικής συνοχής. Επιτρέψτε μου εδώ να εκφράσω την ελπίδα ότι ο δυναμισμός και η δέσμευση της Πολωνικής Προεδρίας είναι πράγματα τα οποία θα κυριαρχήσουν μια που και η Επιτροπή των Περιφερειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ξεκινήσει τη δουλειά της. Όντως, πρόκειται για μια πολιτική επενδύσεων και αυτό θα φανεί και τις επόμενες μέρες. Είναι ένα έξυπνο σχέδιο, συμπεριλαμβάνει όλους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται και τι σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι μόνο και από όλους εσάς, είναι αυτό το οποίο θα κάνει την πολιτική μας μια πολιτική που θα χαίρει εμπιστοσύνη. Όντω πρέπει με φύ τρόπο να ξεκινήσουμε και πάλι να ενισχύουμε την απασχόληση. Και πρέπει να συμμετέχουμε όλοι, ακαδημαϊκοί επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, η πόλεις, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε προσπάθειες υπέρ μιας ανάπτυξης και μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας που θα προσφέρει καλύτερες θέσεις απασχάλησης και καλύτερα, καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε εδώ και θέλω να ζητήσω από την Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών την κυρία Πρέσο και μετά από τον Επίτροπο Χάνης να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Ντανούτα. Και εγώ από πλευράς μου χαιρετίζω τους Προέδρους, την Υπουργό, τους και τις βουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών και όλους τους προσκεκλημένους που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Με μεγάλη μου χαρά, εξ ονόματος της Επιτροπής μου, της Επιτροπής μας μάλλον, κηρύσω την έναρξη αυτής της ένα της εβδομάδας για τις ευρωπαϊκές πόλεις που συμπίπτει και με την ολομέλεια της Επιτροπής Περιφερειών η πολιτική συνοχή. ήταν πάντοτε στο κέντρο των συζητήσεών μας και στα όσα μας απασχολούν στις συναντήσεις αυτές. Φέτος βρισκόμαστε πέντε μέρες μετά την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχετικού νομοθετικού πακέτου. Ευχαριστώ λοιπόν καταρχάς την κυρία Χούμπνερ που με τη στήριξή της επέτρεψε να συναντηθούμε και πάλι εδώ στο ημικύκλιο και ευχαριστώ και τους Προέδρους Μπούζεκ και Μπαρόζο καθώς και την Υπουργό Μπιενκόφσκα για την παρουσία τους και τις παρουσιάσεις που θα κάνουν εντός ολίγου. Στις αρχές του φθινοπόρου 2011 βλέπουμε ότι κάθε μέρα υπάρχουν άσχημες ιδέες για δύο μέτωπα. Τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα προβλήματα με τις νομισματικές αγορές και την, ε, το δημόσιο χρέο, καθώ και τον αποκλεισμό, την ανεργία και τι κοινωνικέ εξέλιξει. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα περισσότερο από ποτέ να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και με τρόπο ισχυρό και σαφή. Αναλαμβάνοντα τι δικέ τη αρμοδιότητε. Ο πρόεδρο Μπαρόζο μα το είπε πολύ ξεκάθαρα και την περασμένη εβδομάδα στο μήνυμά του, το οποίο νομίζω ότι και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου το έχουν καταγράψει καθώς και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της, Ευρωπαϊκής, ε, των Περιφερειών, ε, αποδέχτηκαν το μήνυμα αυτό και θα τον στηρίξουν. Έτσι λοιπόν με τη στρατηγική του 2020 έχει καθοριστεί ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε, αλλά τώρα θα πρέπει να εξευρεθούν και τα απαραίτητα κονδύλια μέχρι και την έγκριση του προπολογισμού. Όπως με την πρόταση για 0,05% του εθνικού ΑΕΠ. Ε, η συνοχή στι τρει διαστάσει, στην κοινωνική, την οικονομική και την εδαφική, θα πρέπει να θεωρείται ω μια πολιτική που μπορεί μόνο πλεονεκτήματα να φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια απαραίτητη προπόθεση ώστε να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητά μας στην οικονομία και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, αλλά και να στηρίξουμε τις, μα δημοκρατίες μας και την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να διστάσουμε να κάνουμε μια διάγνωση του ποιες είναι οι δυσκολίες που περνάει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Με κάθε ειλικρίνεια και θάρρος. Κάποιοι δικαιολογούν την ε, συμπεριφορά αναδίπλωση ορισμένων προ τα εθνικά του συμφέροντα, όμω η Ευρώπη δεν θα υποφέρονται από ένα πλεόνασμα συνοχή, ούτε από μια υπερβολικά γενναιόδορη πολιτική συνοχή. Το αντίθετο είναι θύμα του ότι δίνεται, ε, εντείνονται μάλλον οι κοινωνικέ ε, διαφορές και η έλλειψη ισορροπίας. Και αυτό και μεταξύ των περιφερειών και επαρχιών. Έτσι λοιπόν ο ρόλος μας ως εκπροσώπων των τοπικών αρχών αυτοδιοίκηση είναι να υποδείξουμε την προστιθέμενη αξία τη πολιτική συνοχή. Περισσότερο από κάθε άλλη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η πολιτική επιτρέπει να προβληθεί η αξία τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε επίπεδο περιφερειών για του πολίτε και μπορεί να δώσει και μια κατάλληλη απόκριση, μια συντονισμένη απόκριση στι ανάγκε του και τα προβλήματά του. Είναι η μόνη πολιτική ανάπτυξη και επένδυση η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τι αρνητικέ συνέπειε τη εσωτερική αγορά και να βοηθήσει του περιφερειακού παράγοντε να ε, αδράξουν τι ευκαιρίε που μπορεί να προκύπτουν. Σε μια περίοδο κρίση, λοιπόν, είναι διπλά απαραίτητη η πολιτική αυτή, διότι παρουσιάζει μια ευκαιρία για όλου όσοι επλήγησαν να αλλάξουν την κατάστασή του και να στηριχθούν οι επενδύσει που μέσω πρόθεσμα μπορούν να μα οδηγήσουν σε μια ανάπτυξη ικανοποιητική και σε καινοτόμε λύσει πριν δώσω έμφαση στις διάφορα, στα διάφορα θετικά στοιχεία της πολιτικής συνοχής, να εκφράσω και την απογοήτευσή μου όπως συμβαίνει με τους ε, τάβρους στις ταυρομαχίες όταν τους ε, ε, δείχνουν την, ε, το κόκκινο πανί όταν κουνάνε μπροστά του το κόκκινο πανί. Το ίδιο λοιπόν και με τι οικονομικέ δυσκολίε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ε, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μα διότι η θέση τη Επιτροπή των Περιφερειών παραγνωρίστηκε όπω έγινε και για το Ευρωκοινοβούλιο. Εμεί επαναλάβαμε ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε οι περιφέρειε και οι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση να υποστούν τι ενδεχόμενε συνέπειε τη ανικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων να καλύψουν τι υποχρεώσει του, υποχρεώσει οι οποίε προκύπτουν από το πλαίσιο πλαίσιο τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Σε μια περίοδο κρίση, όπω θα μπορούσε να δικαιολογείται, ε, οι επιχειρηματίε ε, που θα έπρεπε να κάνουν επενδύσει κατά τη ανεργία, που έχουν κάνει προσπάθειε ε, να δώσουν μόρφωση και εκπαίδευση στου νέου με τα δικά του τα κονδύλια. Όλοι αυτοί που προσφέρουν ένα κοινωνικό έργο δεν μπορεί να προστατεύονται λιγότερο σε σχέση με του γεωργού Λογουχάρη ή άλλου πολίτε που λαμβάνουν άμεσε βοήθειε. Ακόμη και αν η τωρινή πρόταση φαίνεται ότι ανοίγει την πόρτα σε μια προσέγγιση συνεργασία. Πιστεύω ωστόσο ότι κατά τι διαπραγματεύσει που πρόκειται να ξεκινήσουν θα πρέπει και εμεί να φροντίσουμε να ακουστεί με ηχηρό τρόπο η δική μα φωνή και άποψη. Θα ήθελα τώρα να περάσω και στα θετικά στοιχεία τα οποία είναι πολλαπλά. Πρώτον, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο το οποίο βασίζεται σε πέντε ταμεία τα οποία κινητοποιούν τι διάφορε πολιτικέ μα πλαίσιο το οποίο αναγγέλει και μας επιτρέπει να προνοιονίζουμε μεγαλύτερη απλούστευση στις ε, τοπικές υλοποιήσεις του. Έπειτα η αναγνώριση της εταιρική σχέσης με τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που ε, επιτρέπει σχέσεις εταιρικής ε, συνεργασίας και συντονισμό. Επίση, οι προσπάθειε απλούστευση που ε, περιέχονται στο στου προτινόμενου κανονισμού είναι καλοδεχούμενε. Επίση, για την εδαφική διάσταση στι συμβάσει εταιρική σχέση μέσω του συντονισμού των πέντε ταμείων θα είναι πολύ χρήσιμα. Όπω και η ενοποιημένη προσέγγιση τη εδαφική ε, ανάπτυξη, ο εντοπισμό ε, των γεωγραφικών περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η ρητή αναγνώριση τη εδαφικότητα, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδυας. Αυτά είναι θετικά στοιχεία. Τέταρτον, η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ε, περιφερειών, των μεταβατικών όπως λέγονται, και πέμπτο, η, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που και αυτό θα στηρίζει την πολιτική συνοχή με την προοπτική ε, κονδυλίων που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένε περιφέρειες. Έκτον, η ενίσχυση τη εδαφική ε, συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με, με ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και αναγνώριση του ρόλου τη στην καινοτομία που μπορεί να προσφέρει και στην ανανέωση τη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Έβδομο θετικό στοιχείο που μπορεί να σα εκπλήξει κιόλα είναι οι, οι εσωτερικέ προποθέσει, οι εσωτερικοί όροι που τίθενται. Δηλαδή, ανάλογα με τις τοπικές αρχές, ε, τις αρχές μάλλον τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μπορεί αυτό να γίνει ένα εργαλείο στα χέρια των κατώμελών για να ελέγχουν εφόσον μπορούν να επιβάλλουν όρους και να βλέπουν ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει η ΜΕΝ και η ΔΕ. Συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι επί παραδείγματι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σημαντικό είναι να στηρίζει προγράμματα τοπικής ένταξης, επαγγελματικής ένταξης ακόμη κι αν η εθνική νομοθεσία μπορεί να έχει διαφορετικές ε, διαθέσεις ή ε, διαφορετικούς κανόνες. Σε αυτήν την προκαταρκτική μου ομιλία δεν είναι δυνατόν να καλύψω ένα τόσο ευρύ πεδίο βεβαίως κυρίες και κύριοι, διότι σήμερα ε, μπροστά σας έχω την μοναδική ευκαιρία να απεικονίσω εν συντομία τις δικές μας θέσεις και να τις ε, κάνω να ακουστούν και στους προέδρους του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και την αρμόδια Υπουργό εκ μέρους της Πολωνικής Προεδρίας για την Περιφερειακή Πολιτική. Το ίδιο και για την Επίτροπο και την Πρόεδρο της Επιτροπής Ρέτζι, της ε, περιφερειακή ανάπτυξη, με τους οποίους θα συνεργαστούμε βεβαίως στενά του ερχόμενου μήνε, ώστε να αποσπάσουμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτές τις προτάσεις. Δεν μπορώ βεβαίω παρά μόνον να επαναλάβω πολύ σύντομα τις θέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών. Ήδη αρχίσαμε να τις επεξεργαζόμαστε και προφανώς στο προσεχές διάστημα τις ερχόμενες εβδομάδες θα τις εγκρίνουμε και επισήμως. Ευχαριστώ λοιπόν όλους, όλες μάλλον τις παρούσες και όλους τους παρόντες για την ε, προσέλευσή τους και ελπίζω οι μέρες αυτές για τις ευρωπαϊκές πόλεις να μας επιτρέψουν να δείξουμε την αξία της εδαφικής πολιτικής και της περιφερειακής διάστασης στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι φίλοι των περιφερειών και των πόλεων και των χωριών της Ευρώπης. Μια και θα έχω τη δυνατότητα υστερότερα πιο διεξοδικά να τοποθετηθώ για την πρώτη πρότασή μας, θα ήθελα απλά εδώ στην αρχή να δραχθώ της ευκαιρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σας χαιρετήσω θερμά και να σας υποδεχθούμε θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω για την δυνατότητα αυτών των ανοιχτών ημερίδων Open Days που κάθε χρόνο όλο και πιο έντονα διεξάγονται σε μεγαλύτερο βάθος είναι η πιο σημαντική συνάντηση για την περιφερειακή πολιτική που γίνεται. Έχουμε φίλους από πολλές άλλες περιφέρειες και περιοχές του κόσμου που μπορούμε να καλοχαιρετήσουμε εδώ 110 σεμινάρια, πάνω από 250 άλλα αποκεντρωμένα θα έλεγα ως πρωτοβουλίες γεγονότα που στις πολιτικές μας στις πόλεις ε, και στο σύνολο της Ένωσης διεξάγονται 25.000 άνθρωποι τις επόμενες ημέρες θα ασχοληθούν σε βάθος με το θέμα του πώς μπορεί κανείς με φιέστερο τρόπο, με πιο αηφόρο τρόπο, με πιο ολοκληρωμένο τρόπο να δράσει για το μέλλον των ευρωπαϊκών περιφερειών και να επενδύσει σε αυτό το μέλλον στις περιφέρειες. Έχουμε μια πρόταση για, για τη ρύθμιση αυτού του πλαισίου που όλα τα τμήματα και τα κομμάτια τα ολοκληρώνει σε ένα ενιαίο σύνολο. Θέλω να ευχαριστήσω για την μ, πολύ θετική αντίδραση και τοποθετήσεις θετικές στην πρότασή μας. Υπάρχει το ένα ή άλλο θέμα που τους επόμενους μήνες θα πρέπει να συζητηθεί και πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί. Το αναμέναμε αυτό και είναι φυσιολογικό και ομαλό. Μια σύντομη αξιολόγηση που μια και τις τελευταίες ημέρες ρίμνησε για πολύ θόρυβο η μακροοικονομική όρη και προϋποθέσεις έχουμε μια ξεχωριστή δυναμική όσον αφορά την οικονομική κρίση και τις οικονομικές εξελίξεις. Το είδαμε αυτό ως γεγονός και πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το γεγονός. Και γι' αυτό πάντα το αίτημα η διεκδίκηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο και έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δραστηριοποιηθεί, να αντιδράσει και όταν είναι αναγκαίο να υιοθετήσει μηχανισμούς κυρώσεων που πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να δράσει αποτελεσματικά. Όταν υποβάλουμε μια τέτοια πρόταση πρέπει φυσικά να συζητήσουμε συζητηθεί αυτή και θα συζητηθεί. Αλλά η αρχή αυτή πρέπει να είναι δεδομένη. Ότι όταν δηλαδή κράτη-μέλη <clears throat> με την δυνατότητα να παρέμβουν όταν έχουμε θέματα μακροοικονομικών συνιστοσών, όλες οι προτάσεις, όλα τα αιτήματα όταν αγνοούνται και παραμελούνται, τότε θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. Και αυτό είναι το πνεύμα αυτής της πρότασης. Με ευφυή τρόπο θα πρέπει να συζητήσουμε χωρίς να αναβάλουμε το θέμα, θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και τις επόμενες ημέρες να συζητήσουμε για όλες τις άλλες πτυχές και παραμέτρους της περιφερειακής πολιτικής που θα συνεισφέρουν στο τέλος τέλος στην αηφορία αυτής της ε, περιφερειακής πολιτικής. Από μια φιλανθρωπική charity πολιτική να γίνει μια πολιτική επενδύσεων που θα ενεργοποιήσει τις περιφέρειες και τους ανθρώπους ώστε να υπάρχει πρόσθετη ευρωπαϊκή αξία που θα δημιουργηθεί. Αυτό είναι το πνεύμα των κανονισμών και των ρυθμίσεων που προτείναμε και υποβάλαμε και χαιρόμαστε για την ζωντανή συζήτηση που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Σας εύχομαι καλή δουλειά στις συζητήσει σας. Ευχαριστώ. Uh, Θέλω τώρα να προχωρήσουμε στους επόμενους ομιλητές μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Πούτσεκ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για τις παρουσιάσεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ εμείς οι ευρωβουλευτές που σας φιλοξενούμε εδώ. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο φόρουμ που υπάρχει όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη σε ολόκληρο το κόσμο. Είναι οι δικές σας ημερίδες λοιπόν, αλλά είναι και η δικιά μας ευρωπαϊκή ημερίδα, μια που βρισκόσαστε εσείς εδώ σε μας. Θέλω να υπογραμμίσω ένα πράγμα που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό από πλευρά και δικιά μου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι ότι πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες μας. Ιδιαίτερα μάλιστα τώρα. Και αυτό γιατί οι καιροί δεν είναι εύκολοι. Κυρίως για τους πολίτες μας. Και εσείς εκπροσωπείτε την τοπική και περιφερειακή κοινότητα. Άρα εσείς βρίσκεστε κοντά στους πολίτες μας και εσείς μπορείτε να τους επηρεάσετε, μπορείτε να τους εξηγήσετε τι πραγματικά κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη στήριξή σας, χρειαζόμαστε τις συμβουλές σας, χρειαζόμαστε τη δράση σας. Χωρίς τη δικιά σας δράση, επιτρέψτε μου να το υπογραμμίσω αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες. Τώρα όμως είμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο. Γι' αυτό και πρέπει να συνεργαστούμε οι πολιτικοί μεταξύ μας πολύ περισσότερο, πολύ πιο συχνά, προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για τους πολίτες μας. Και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να πετύχουμε, χάρη σε εσά πρώτα απ' όλα. Έχω εδώ ετοιμάσει κάποιες σημειώσεις για τη σύντομη ομιλία μου, αλλά είναι στα πολωνικά, στη μητρική μου γλώσσα, οπότε θα συνεχίσω στα πολωνικά διότι δεν μου είναι πολύ εύκολο να μιλήσω άλλη γλώσσα. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Είναι τεράστια σημασία. εμείς να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να κατανοήσουν οι πολίτες περί τίνος πρόκειται. Είναι μείζον εγχείρημα αυτό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας. Πρέπει να υιοθετήσουμε νομοθετικό έργο, να, να νομοθετήσουμε με όριμο τρόπο για τα θέματα που αφορούν την Ήπειρό μας σε αυτή τη συνιστόσα και κάνοντας αυτό πρέπει να είμαστε κατανοητοί για τους πολίτες μας. Όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, ήδη διεξάγονται συζητήσεις για νομοθετικές προτάσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τα τελευταία δύο χρόνια <clears throat> είδαμε το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Ο Επίτροπος Χάν θα επισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα όμως εγώ να αναφέρω ότι πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις από κοινού. Το Συμβούλιο, οι Υπουργοί των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να συνομοθετούμε. Είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Από κοινού είμαστε συναρμόδιοι η συνάντηση των Υπουργών των Κρατών Μελών, οι κυβερνήσει των Κρατών Μελών στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είμαστε συναρμόδιοι. Έχουμε Πλήρει αρμοδιότητες και ευθύνε ως Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι τόσο συμβολικό και σημαντικό το ότι συνερχόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ακούσουμε τις απόψει σας για αυτά τα θέματα. Είναι ζωτική σημασία, καθώς θα λαμβάνουμε αποφάσεις για θέματα που αφορούν τις τοπικές αρχές και τι περιφερειακέ αρχέ να μπορούμε να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε την σημασία των δημοσιονομικών θέμα, θεμάτων και του προϋπολογισμού. Θέλουμε να διαθέσουμε για όλους τους πολίτες μας, για τις τοπικές αρχές, για τις επιχειρήσεις, τα αναγκαία πλαίσια. Κατανοούμε από πού προέρχεται η πίεση να υπάρχουν εξοικονομήσεις και περικοπές. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι πολύ αξιόλογο, πολύ σημαντικό. Το να περικοπεί, να συρρυκνωθεί θα μπορούσε να έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Καλωσορίζω την παρουσία του Ζωζέ Μανουέλ Ντουραν Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ καλό είναι ότι παρήσαστε κύριε Μπαρόζο, διότι ο προπολογισμό που προανέφερα σημαντικά προσχεδιάζεται και καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι στα χέρια της. Το Συμβούλιο και το ε, Κοινοβούλιο συνδιαβουλεύονται και διαπραγματεύονται. Όμως εδώ υπάρχει πολύ σημαντικός ρόλος. Ο πολιτισμό έχει τεράστια σημασία, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της περιφερειακής πολιτικής. Και είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε από τον πρόεδρο Μπαρόζο τα σχετικά. Είναι πολύ σημαντικό για την στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Και αυτή η στρατηγική γεννήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πατέρας της εντό εισαγωγικών, ο γονιός της είναι ο Ζωζέ Μανουέλ Ντουράν Μπαρόζο. Εκείνο είναι ο δημιουργό αυτής της στρατηγικής. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε χρονικά αυτή την συνιστόσα. Θα γνωρίζετε κυρίες και κύριοι περί τίνος πρόκειται για την στρατηγική για το 2020. Είναι το να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι το να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Είναι το να προαγάγουμε την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες μας. Αυτές οι δουλειές, οι θέσεις απασχόλησης στο τέλος, τέλος είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Γι' αυτό έτσι καθώς θα λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας σχετικά θα πρέπει να διαπιστώσουμε πού βρίσκονται τα πιο ευάλωτα σημεία μας. Χαμηλή παραγωγικότητα, υψηλά επίπεδα δημόσιας υπερχρέωσης, φραγμοί και προσκόμματα όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά. Επιτρέψτε μου να σας επεξηγήσω κυρίες και κύριοι γιατί και πώς τοποθετούμε για αυτά τα θέματα. <clears throat> Λίγο πιο μακριά μια κοινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση διεξάγεται την παρουσία του Επιτρόπου Μπάρνιε για την εσωτερική αγορά υπάρχουν εκπρόσωποι 18 κρατών μελών που συνέρχονται. Φυσικά υπάρχουν και ευρωβουλευτές. Η Πολωνική Προεδρία επίσης εκπροσωπείται περί τίνος διαβουλεύονται. Συζητούν και διαβουλεύονται για να βρουν τρόπους να ολοκληρωθεί η ενιαία εσωτερική αγορά, να βρουν τρόπους να λειτουργήσει πιο σωστά και πληρέστερα η ενιαία εσωτερική αγορά. Και υπάρχει εκεί ένας δεσμός και ένας κρίκος που μας συνδέει με την περιφερική ανάπτυξη. Αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε την οικονομία πρέπει να δράσουμε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Και το λέω αυτό για να καταστήσει σαφές ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε πολλά πράγματα σε εξέλιξη που αλληλοεπικαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται και που αν όλα αυτά δράσουν συνολικά μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε διέξοδο από την κρίση. Εν κατακλείδη επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια κυρίες και κύριοι γιατί αυτός ο προϋπολογισμός έχει τέτοια μεγάλη σπουδαιότητα επειδή βοηθάει όλες τις χώρες μας χωρίς καμιά εξαίρεση να επιτύχουν την ανάπτυξη, επειδή είναι, έχει μοχλική επίπτωση, είναι ένας μοχλός οικονομικής δράσης και αποτελεσματικότητας. Μοχλικά μας επιτρέπει να δράσουμε και να κινητοποιήσουμε πολύ περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη από ότι μόνος του ο προϋπολογισμός θα μπορούσε να πετύχει. Επίσης αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και μειώνεται η ανεργία. Δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και επίσης ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει και προ περιέχει έχει προνοήσει για την χρηματοδότηση της καινοτομίας και της έρευνας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα μπορούσε κανείς να είναι καινοτόμος και αποτελεσματικός χωρίς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη. Πάλι εδώ υπάρχει σύνδεσμος και συνάρτηση με την περιφερική ανάπτυξη, διότι προς αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να κινηθούμε. Και φυσικά στο τέλος τέλος αυτή είναι μια πολιτική που απέδειξε την αξία της και κατέδειξε την αξία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εδώ και πολλά χρόνια στρατηγική, πολιτική του να επενδύουμε στις περιφέρειες. Επενδύοντας στις περιφέρειες μπορούμε να επενδύσουμε στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η περιφερειακή πολιτική πρέπει να έχει προτεραιότητα και τον σωστό το σωστό μέρος και τόπο που πρέπει να λαμβάνει στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι με κάθε στένος και αποφασιστικότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει πολιτικές υπέρ της συνοχής και υπέρ της περιφερικής ανάπτυξης και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που έχει τέτοια σημασία για εκατομμύρια ανθρώπους που είτε έχασαν τη θέση απασχόλησης εργασίας τους είτε ψάχνουν να βρουν μια νέα εργασία, μια νέα θέση απασχόλησης πώληση στην ευρωπαϊκή αγορά. Στεναρή λοιπόν υποστήριξη, στεναρή αποφασισμένη αποφασιστικότητα στην υποστήριξη που παρέχουμε. Αυτό σημαίνει ότι πάντα υποστηρίζουμε νέες προτάσεις και νέες λύσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο εκ του αναζητούμε και αποζητούμε την δική σας υποστήριξη ως εκπροσώπων της περιφερειακής και τοπικής κοινωνίας. Είμαι πεισμένος ότι αυτοί, οι, αυτές οι ημερίδες θα μας βοηθήσουν προς αυτό το στόχο. Είναι το μεγαλύτερο φόρουμ, η μεγαλύτερη πλατφόρμα για την περιφερειακή ανάπτυξη στην οικουμένη και σίγουρα θα δράσει με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, για τα θερετικά σας λόγια. Τώρα, καλώ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ζωζέ Μανουέλ Παρόσο, για την ε, δικιά του παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ Τζέρσι Μπούσικ, αγαπητή Υπουργέ που εκπροσωπείται εδώ την Πολωνική Προεδρία, κυρία Πρόεδρε της ε, Επιτροπής των Περιφερειών, κυρία Μπρέσο, αγαπητή Πρόεδρο της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Περιφέρειες, κυρία Χούμπνερ, κύριε Χάν, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι εκπρόσωποι των περιφερειών, των πόλεων και των, δήμων, μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να συμμετέχω εδώ στις ένατες ημερίδες που θεωρώ ότι έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν. Είναι πραγματικά μια σημαντική στιγμή για την Ευρώπη. Είναι η στιγμή όπου μαζί ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και περιφέρειες χτίζουμε το μέλλον. Με εκπλήσει επίση, το γεγονό ότι σα βλέπω εδώ τόσο πολλοί αριθμού και από τόσο διαφορετικές γωνιές της Ευρώπη να αγωνίζεστε υπέρ τη πολιτική μα συνοχή, αλλά και υπέρ τη ίδια της Ευρώπη. Για μένα αυτή η αλληλεγγύη, κατεξοχήν αλληλεγγύη είναι η πολιτική συνοχή, είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι έχουν αποφελωθούν από αυτή. Δεν είναι μόνο μια πολιτική σύγκληση, είναι και μια πολιτική όμως ανάπτυξης που δημιουργεί απασχόληση δημιούργησε πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις απασχόληση τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι μια πολιτική που επενδύει στην ε, μόρφωση, επενδύει και στις υποδομές. Είναι μια πολιτική που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάνω από 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι λοιπόν η πολιτική συνοχής και βοηθάει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες τις πιο αδύναμες οικονομικά έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν, αλλά επιτρέπει και σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλες τις περιφέρειες να βρουν καλύτερα τη θέση τους μέσα στην εσωτερική αγορά. Πρόκειται δηλαδή για μια αλληλεγγύη, αλλά πρόκειται και για μια πολιτική ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση σε ολόκληρη την ιστορία της, γιατί νομίζω ότι ζούμε τις πιο ε, λεπτές, τις πιο δύσκολε στιγμές από τότε που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει σήμερα όσο ποτέ να ενωθούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν πάνω απ' όλα είναι περισσότερη ε, συνοχή, περισσότερη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Ναι, αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι μεγαλύτερη συνέπεια από τις πολιτικές μας και μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στην πολιτική μας ε, συνοχής, την πολιτική ανάπτυξη, στην πολιτική μας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στη στρατηγική μας δηλαδή για το 2020. Όπως ε, το έλεγα και στις 27 Σεπτεμβρίου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόνο ενωμένοι μπορούμε να βγούμε από την οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική κρίση που διανύουμε. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου για να βρούμε λύσεις και να τις βρούμε αυτές τις λύσεις και να τις εφαρμόσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Μέσα σε αυτήν λοιπόν την τόσο απαιτητική περίοδο θέλω να ευχαριστήσω τις, για τις προσπάθειές τους που έχουν κάνει τοπικές και περιφερειακές αυτοδικήσεις. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η δέσμευση των περιφερειών και των πόλεων είναι κάτι αναγκαίο, πραγματικά αναγκαίο, προκειμένου μαζί να μπορέσουμε να χτίσουμε μία ένωση σταθερότητας και ευθύνη, μία ένωση ανάπτυξης και αλληλεγγύης. Δεν μπορεί να υπάρχει σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να έχουμε σταθερότητα στι περιφερειέ μα. Δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στι περιφερειέ μα. Και ούτε μπορεί να υπάρχει μια δυνατή ένωση χωρί αυτά τα δύο στοιχεία. Την αλληλεγγύη δηλαδή από τη μία και την υπευθυνότητα από την άλλη. Μία ένωση σταθερότητας και ευθύνη είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις και για να προετοιμάσει το μέλλον. Και γι' αυτό ακριβώς οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από τους ηγέτες ε, κρατών ε, και κυβερνήσεων στην ε, προηγούμενη διάσκεψη κορφής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν αυτή η μεταρρύθμιση θα έχει επικυρωθεί από όλου, η συμφωνία τη 21η Ιουλίου, όταν λοιπόν θα έχει επικυρωθεί από όλου η συμφωνία αυτή, τότε θα μπορέσει ο μηχανισμό να χρησιμεύσει για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, αλλά και για να ενισχύσει τι παράγωγε αγορέ και να βοηθήσει να αποφύγουμε ε, να ε, επεκταθεί περισσότερο η κρίση. Τα, το τελευταίο διάστημα εγκρίθηκε και το πακέτο των έξι συμφωνιών που ενισχύει τη σταθερότητα και ενισχύει και τις μακροοικονομικές ισορροπίες. Τώρα έχουμε ένα ε, μείγμα το οποίο είναι αναγκαίο και απαραίτητο για την Ευρώπη να ξέρετε ότι αν δεν ξεπεραστεί η κρίση αυτή στην Ευρώπη δεν θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη που χρειαζόμαστε για ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρωζώνης δηλαδή. Οπότε τώρα μετά από τη συμφωνία του Σεπτεμβρίου μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη πριν να ληφθούν οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι περιφέρειες συνδέονται άμεσα. Άρα το σύμφωνο που είναι σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνει και τις περιφέρειές σας. Ναι, τα μέτρα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν φτάνουν. Και γι' αυτό όταν μίλησα για την κατάσταση στην Ένωση, ζήτησα να θέσουμε σε εφαρμογή έναν οδικό χάρτη για μια πιο φιλόδοξη Ευρώπη, που ανταποκρίνεται μέσα σε ένα κοινοτικό πλαίσιο στις διάφορες προκλήσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Η κατάσταση στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα το πιο επίγον αυτή τη στιγμή, αλλά επίσης είναι και η πρόληψη του κινδύνου διάδοσης και επέκτασης της κρίσης. Επέκτασης είτε στο δημόσιο χρέος, είτε στο τραπεζικό και δημοσιονομικό σύστημα αλλού. Η πολιτική ανάπτυξη, έπειτα, γιατί είπαμε, χρειάζεται σταθερότητα. Αλλά τις προσπάθειες για σταθερότητα πρέπει να τις συνοδεύσουμε και προσπάθειες ανάπτυξης προλαμβάνοντας την κατάσταση και προβλέποντας μέτρα ανάπτυξης. Επίσης χρειάζεται και μια ενισχυμένη διακυβέρνηση μέσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ακριβώ είναι που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι προφανές κυρίες και κύριοι ότι όλες οι προσπάθειες που κάνουμε για να έχουμε περισσότερη πειθαρχία και σταθερότητα δεν έχουν νόημα παρά μόνο αν συνοδεύονται από προσπάθειες για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ανάπτυξη που θέλουμε να είναι βιώσιμη, να είναι δίκαια, και να δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να δει πώς ε, θα φροντίσει να υπάρξουν μέτρα διαρθρωτικά. Οπότε στην περίπτωση της Ελλάδας εγώ ανέλαβα την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια task force η οποία θα επιτεχύνει την απορρόφηση των διαρθρωτικών ε, κονδυλίων. Πρόκειται για 15 δις ευρώ για την Ελλάδα και μόνο με προγράμματα τα οποία θα ενισφέρουν στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στη χώρα αυτή. Και γι' αυτό και προτείναμε νέους κανόνες συγχρηματοδότησης για τις χώρες οι οποίες ε, χαίρουν μακροοικονομικής ε, αρρωγής. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα εγκρίνουν σύντομα τις προτάσεις μας αυτές. Όλα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι η πολιτική συνοχή και τα διαφορετικά ταμεία είναι σήμερα περισσότερο σημαντικά από ποτέ για να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που με τη σειρά της δημιουργεί απασχόληση για τους νέους πρώτα απ' όλα Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με τεράστια ανεργία, που σε μερικές χώρες η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Πρόκειται για τους δικούς μας νέους, οι οποίοι δεν έχουν πια εμπιστοσύνη στο μέλλον τους. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις. Μια οικονομική ανάκαμψη χωρίς δημιουργία απασχόλησης δεν έχει και πολύ νόημα. Η κρίση δεν πρόκειται να τελειώσει όσο δεν έχει καταπολεμηθεί η ανεργία, όσο δεν έχει μειωθεί δηλαδή σημαντικά η ανεργία στην Ευρώπη. Αυτό επίση που θέλουμε είναι μεγαλύτερη ισότητα. Τη στιγμή που ζητάμε θυσίε από του πολίτε μα είναι σημαντικό να καταλάβουν αυτοί ότι όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τέτοιε θυσίε. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα έκανε μια πρόταση φορολόγηση των δημοσιονομικών συναλλαγών. Πρέπει και ο οικονομικό τομέα να αναλάβει τι δικέ του ευθύνε. Είναι ένα βασικό σημείο για να υπάρχει ισότητα και να υπάρχει εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Κυρίε και κύριοι, η στρατηγική μας για το 2020 κάνει ένα μεγάλο βήμα για να πετύχουμε μια ανάπτυξη βιώσιμη και φύγη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που οι περιφέρειες, οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, ε, συμφωνούν με τους στόχους αυτούς της στρατηγικής μας και είναι προπόθεση για να πετύχει η Ευρώπη του 2020. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς να κινείται. Πρέπει και εμείς να εξελιχθούμε και να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής απομονωμένα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις που έχει οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σημαντικές αλλαγές για να εξυγχρονίσουμε μαζί την πολιτική συνοχής μας. Οι αρχές είναι ίδιες. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξυγχρονίσουμε κάποια από τα μέσα που χρησιμοποιούμε στην πολιτική μα αυτή. Για παράδειγμα, την περιφερειακή πολιτική πρέπει να τη δούμε γενικότερα βάσει των στόχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση για την, το επόμενο πολιτέ ε, πλαίσιο. Πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν θα είναι πιο εύκολη η συζήτηση που θα γίνει από τη συζήτηση για τον επόμενο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πιο δύσκολη στιγμή για να συζητάει κανείς για πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση των προπολογισμών των περισσότερων χωρών μας. Άρα πρέπει να εξηγήσουμε για την Ευρώπη, πρέπει να εξηγήσουμε γιατί ένα ευρώ το οποίο δαπανάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει περισσότερο νόημα από ένα ευρώ το οποίο δαπανάται σε εθνικό επίπεδο. Και αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και εθνική στήριξη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια, αλλά και από τα κοινοβούλια των χωρών μελών μας, από όλες τις χώρες ε, μέλη, γιατί χρειάζεται ομοφωνία των κρατών μελών. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε από πιο κοντά την πολιτική συνοχής στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και σε σχέση επίση και με το σύμφωνο σταθερότητα. Και πρέπει να πάρουμε μαθήματα από το παρελθόν. Ξέρουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο μακριά όσον αφορά το συντονισμό τη δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών. Προσπαθούμε να έχουμε μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετικέ πολιτικέ στι διάφορε χώρε. Αν θέλουμε να έχουμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, πρέπει να συνδέονται οι πολιτικέ μα μεταξύ του. Η πρότασή μας πιστεύουμε ότι είναι σωστή και ισορροπημένη. Σταδιακά θα προχωρήσουμε και θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση από την οποία όλοι έχουν να κερδίσουν. Μοιρασμένη ευθύνη με στόχο να διασφαλίσουμε ότι η αποτελεσματικότητα των δαπανών μας δεν υπονομεύεται από ε, μη υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές. Γιατί τότε είναι πολύ αργά. Τη πολιτική συνοχή μας θέλουμε να τη βασίσουμε στη συνυπευθυνότητα και στην αλληλεγγύη με καλές επιδόσεις και καλά αποτελέσματα. Ο κοινοτικό προπολογισμό και ιδίω τα διορθωτικά ταμεία, όλα τα διορθωτικά ταμεία πρέπει και θα είναι στο, στην πρώτη γραμμή. Θα παρακολουθούμε κάθε ευρώ που θα πανάτε. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να οδηγεί σε ανάπτυξη πολιτικής συνοχής μας. Γι' αυτό ακριβώς, παρόλο που συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά τις πιο δύναμες ε, περιφέρειες, χρόνος προτείνουμε να δημιουργηθεί μια νέα ε, κατηγορία μεταβατικών περιφερειών, η οποία θα καλύπτει τις περιφέρειες εκείνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, των οποίων το επίπεδο μειώνεται και όπου θα βρίσκεται ανάμεσα στο 75% και το 90% του μεσουόρου. Πολλά έχουν συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ήταν προφανέ να καταλήξουμε σε αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο να διασφαλίσουμε το μέλλον τη περιφερειακή πολιτική μα και τη πολιτική συνοχή. Γιατί αυτέ οι δύο πολιτικέ δεν είναι για να βοηθήσουμε μόνο τους πιο δύναμους αλλά είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική που έχει νόημα για να πετύχουμε τη συνοχή, για να πετύχουμε την αλληλεγγύη, αλλά και για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε τη στήριξη των κρατών μελών, γιατί τη χρειαζόμαστε για να πετύχουν οι στόχοι μας και να έχουμε έτσι μια πιο φιλόδοξη περιφερειακή πολιτική. Πρέπει να επενδύουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε όσον αφορά το κεφάλαιο. Και το ποιο κεφάλαιο είναι αυτό, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και προτείνουμε ο ρόλος του κοινωνικού ταμείου να ενισχυθεί για να στηρίξει την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την ε, παιδεία και την κατάρτιση γενικότερα. Θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία προς όφελος ε, του Ταμείου Συνεχής, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με δικιά μου πρωτοβουλία μάλιστα αποφασίσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή που δέχτηκαν και αποφάσισαν καινούς κανόνες για όλους τους χώρους συνεργασίας όσον αφορά τα διάφορα κονδύλια μας. Έτσι απλοποιείται το μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εξυγχρονισμένη πολιτική που να λαμβάνει υπόψη την αγωνιστικότητα, μια πολιτική συνοχής δηλαδή που να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικότητας και της υπεύθυνη αλληλεγγύης. Και θέλω να τελειώσω με μια έκκληση, ειλικρινή έκκληση, μετά τα όσα είπε και ο πρόεδρος Μπούζεκ. Ζούμε μέσα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και εσείς ως Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξετε την Ευρώπη στις περιφερειές σας και στις χώρες σας. Είναι πολύ σημαντικό οι περιφέρειες της Ευρώπης να πούν στις κυβερνήσεις και στις ε, προ... διάφορες πρωτεύουσέ σας πόσο σημαντική είναι αυτή η περιφερειακή μας πολιτική, ότι τα χρήματά της δεν είναι χρήματα για τις Βρυξέλλες, αλλά είναι χρήματα για τις περιφέρειες της Ευρώπης, για τους εργαζόμενους της Ευρώπης, για τους αγρότες, για όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα μέλλον στην Ευρώπη για τους πολίτες της Ευρώπης, για αυτούς που είναι στην ανεργία ή για αυτούς που φοβούνται ότι θα καταλήξουν στην ανεργία. Είναι μια επένδυση λοιπόν στο μέλλον της Ευρώπης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτή δηλαδή την συνενοχή κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ευρωπαϊκές ε, περιφέρειες. Και αυτή την έκκληση θέλω να κάνω σε εσά για να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και εσείς να τους εξηγήσετε ότι δεν υπάρχει καμία υπερβολή όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία υπερβολή συνοχή στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία υπερβολή Ευρώπη. Αντίθετα, αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη είναι περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη υπευθυνότητα. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε, που υπήρξατε τόσο σαφής όσο σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και την περιφερειακή της πολιτική. Τώρα, εκ μέρους της Πολωνικής Προεδρίας, να προσκαλέσω την κυρία Ελσμπιέτα Μπιενκόφσκα να μας μιλήσει και εκείνη για το πού βρισκόμαστε σε εξής την πολιτική αυτή για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, Κύριε Ευρωβουλευτέ, κύριε Εκπρόσωπο, είναι μεγάλο προνόμιο για μένα να μπορώ να παρακολουθήσω αυτές τι εργασίε, αυτής τη ολομέλεια που ξεκινούν τις ένατες ημερίδε. Είχα συμμετάσχει, είχα εμπλακεί σε αυτές τις συναντήσεις επί πολλά χρόνια ω εκπρόσωπο μιας περιφέρειας τη Πολωνία. και τα τελευταία χρόνια ω υπουργό για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Πολωνία. Οι σημερινές, οι εφετινές εκδηλώσεις διεξάγονται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Είναι ιδιαίτερη συγκυρία για τις συζητήσεις για τα δημοσιονομικά, για τον μελλοντικό προϋπολογισμό, για τις μελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ειδικού χαρακτήρα επειδή αλλάζει ο ρόλος ε, των ευρωπαϊκών πόλεων ε, και των ε, περιφερειών για την επίτευξη των στόχων μας με την δημοσίευση των κανόνων και κανονισμών όσον αφορά την Πολιτική συνοχή από το 2014 και επέκεινα και εφεξίσα Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Πολωνική Προεδρία ξεκίνησε τις συζητήσεις επ' αυτών. Ανέμενε η Πολωνική Προεδρία αυτές τις εξελίξεις, αυτά τα γεγονότα και αδειμονούσε με ιδιαίτερο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα, αυτές οι προτάσεις είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών διαβουλεύσεων και συζητήσεων μεταξύ και της τρέχουσας, της προηγούμενης, των προηγουμένων προεδριών, της προηγούμενης προεδρίας και ιδιαίτερα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κληρονομήσαμε τα προϊόντα, τα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων και θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως βάση, ως θεμέλια για το μελλοντικό μας έργο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Επίτροπο Χάν για την παρουσίαση αυτών των προτάσεων που πολυσχηδώς ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των κρατών μελών. Και αυτέ οι προσδοκίε είναι σαφείς η πολιτική συνοχής θα πρέπει να ενδυναμωμένα να συνδέεται και να συναρτάται με την πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και την συνοχή. Θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικές στρατηγικές που θα σχεδιάζονται για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Παραδοσιακά οι διαπραγματεύσεις οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής, οι διαβουλεύσεις ε, γίνονται σε ομάδες εργασίας ε, για τις διαθωτικές πολιτικές και τα διαθωτικά ταμεία αύριο. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα συζητήσει τις νομικές αυτές τις νομοθετικές προτάσεις. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις και στις ομάδες εργασίας. Το χρονοδιάγραμμα για αυτές τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα στενό οι τριμερείς, δηλαδή Πολωνία, Δανία, Κύπρος από πλευράς Προεδρίας θα ήθελαν να ακολουθηθεί ένας γοργός ρυθμός ώστε μια συμφωνία στο πακέτο να μπορέσει να, επιτευχθεί, να επιτευχθεί μόλις θα υπάρξει ένας συμβιβασμός που θα έχει υιοθετηθεί με βάση τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα έπρεπε να είναι κοινός στόχος όλων μας να καταφέρουμε οι πολιτικές αυτές να λειτουργούν κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, έγκαιρα δηλαδή μέχρι τότε. Είναι Οκτώβριος 2011 τώρα και η Πολωνική Προεδρία έχει δύο μήνες για να, να μπορέσει να παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις. Οι συμφωνίες θα επιτεθούν σε μεγάλο βαθμό δηλαδή υπό την Δανέζικη Προεδρία και υπό την Κυπριακή Προεδρία μελλοντικά. Στόχος μας όμως είναι να προωθήσουμε αυτό το έργο και να το προαγάγουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά και να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε και να προλυάνουμε συμβιβασμούς με τέτοιο τρόπο ώστε να επιλεγούν τα θεματολογικά, τα, οι θεματολογικές μονάδες που θα, θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν το δυνατόν γοργότερα. Ένα από αυτά αυτά τα θεματολογικά θέματα είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Ένας άλλος είναι οι όροι και προϋποθέσεις, ένας άλλος είναι η περιφερική χωροταξία και όλα τα θέματα της περιφερικής συνεργασίας. Πριν από το τέλος, πριν εκπνεύσει η Πολωνική Προεδρία, στοχεύουμε στο να υποβάλουμε έκθεση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Επίσης θα θέλαμε να, είχαμε, να έχουμε μια συνάντηση από πλευράς Υπουργών Γενικών Υποθέσεων ώστε να συνέρθουν οι αρμόδιοι υπουργοί, οι συναρμόδιοι υπουργοί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να συζητήσουν τα κυριότερα στρατηγικά θέματα και τα κυριότερα πιο επίμαχα θέματα που θα έχουν εντοπιστεί από τις ε, ε, συνόδους των ομάδων εργασίας. Ένα από τα ερωτήματα που διατυπώνουμε και διαρωτόμαστε και εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό είναι ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν τα αστικά κέντρα, οι πόλεις, τα κέντρα μας να διαδραματίσουν στις διαπραγματεύσεις και πώς οι απόψεις τους θα μεταφραστούν όσον αφορά το μέλλον της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή. Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω σε αυτό το φόρουμ. Ένας από τους στόχου της Πολωνικής Προεδρίας είναι και παραμένει η ενδυνάμωση, η ενίσχυση της περιφερειακής φιλοδοξίας ο συνιστό σα, στην πολιτική συνοχή ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτόμαστε σε ευρύτερου όρου και προϋποθέσεις για αυτή τη στρατηγική. Έχουμε υπόψη ένα πολύ ευρύτερο φάσμα αυτής της ε, δράσης ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια ως συγκυρία, την χρηματοοικονομική κρίση, την κρίση γενικότερα, μας κατέδειξαν όλα αυτά ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και να εστιαστούμε με ιδιαίτερο τρόπο σε συγκεκριμένους τομείς και άξονες, τις ανάγκες που υπάρχουν εκεί, το δυναμικό και την εμπειρία μας, την πείρα μα. Πρέπει να αποφύγουμε την διαπεδωτική προσέγγιση μιας λύσης για όλα. Και έτσι θα πρέπει σε αυτό το στόχο να δώσουμε τα σωστά αποτελέσματα. Δηλαδή, ενσωματωμένη, ολοκληρωμένη επένδυση, επενδύσεις στο ε, περιφερειακό σκέλος. Η πανοπλία αυτή των μέσων στη φαρέτρα μας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να προαγάγουμε και τα αστικά μας κέντρα. Από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα και στη συνέχεια μέχρι το Δεκέμβριο η Πολωνική Προεδρία έχει ε, φιλοξενήσει και θα συνεχίσει να προγάγει σεμινάρια, διαβουλεύσεις, συναντήσεις όπου αυτά τα θέματα θα εξετάζονται σε πολύ μεγαλύτερο βάθος και λεπτομέρειες από εκπροσώπους των κρατών μελών, από εκπροσώπους των περιφερειακών και τοπικών αρχών όπως επίσης και από εμάς που συμπεριλαμβάνεστε σε αυτόν τον κύκλο. Πάμπολες λοιπόν διαβουλεύσεις ε, και συζητήσεις, όπως εκείνες για την υλοποίηση της ε, στρατηγικής δράσης για την περιφερειακή ανάπτυξη για το 2020 από πλευρά της Ευρώπης, όπως ε, προήχθηκε από την Ουγγρική Προεδρία. Έχουν συζητηθεί θέματα της περιφερειακής συνιστώσας, βιώσιμα αηφόρα μέσα για αυτήν την περιφερειακή διάταξη και συνιστόσα, ενδυναμώνοντας την τοπική διάσταση, την περιφερειακή διάσταση και είχαμε και μία διάσκεψη στη Βασοβία πριν από δύο ε, εβδομάδες ε, για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτή τη συνιστόσα στα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεύτερον, καλύτερος και μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ ομάδων εργασίας που αφορούν ε, τα περιφερειακά θέματα και τα θέματα αστικών κέντρων. Εθνική και ε, διαμεσολαβητές, ε, ομάδες που θα μπορούν να έχουν διαμεσολαβητικό ρόλο, ομάδες εργασίας για την ε, χωροταξική συνεργασία και συντονισμό τρίτων το μέλλον των μέσων και εργαλείων όπως το Epson και το Urban. Ήδη αρκετά πολλά επιχειρήματα έχουν ακουστεί και έχουν αποκαλυφθεί ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν αυτές οι δράσεις, αυτά τα προγράμματα, αυτά τα μέσα. Και μετά η δικτύωση των ευρωπαϊκών πόλεων και ε, πολισμάτων. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε υπό την αιγίδα της Προεδρίας σε αυτό το έργο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη και την πρόοδο των αστικών κέντρων και των πόλεων. Θα έχουμε και τον Οκτώβριο μια διάσκεψη στην Πολωνία, στη Βαρσοβία για αποτελεσματικά μέτρα περιφερικής ανάπτυξης και σε ένα μήνα στις 24 Νοεμβρίου στο Πόσνάνια θα έχουμε μια υψηλού επίπεδου διάσκεψη που θα αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων και των πόλεων όπου θα έχουμε την χαρά να έχουμε εκπροσώπους ε, της Επιτροπής Περιφερειών, των Συμβουλίων Τοπικών ε, Αρχών και Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς επίσης και τους εκπροσώπους που θα συμμετέχουν από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αναμένεται και προσδοκάται ότι θα διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στις συζητήσεις για το μέλλον ε, της πολιτικής συνοχής θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν τη δική σας φωνή, τις δικές σας απόψεις, να ακούσουμε τις απόψεις των εκπροσώπων των πολιτών και μια συνάντηση σαν αυτή είναι ιδανική για να ακουστούν τέτοιες απόψεις. Τίνουμε σε Ευχαριστώ. E, σας ευχαριστώ πολύ Υπουργέ και ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο Συζήτηση και τη συνάντησή μας. Ευχαριστώ τους τρεις προέδρους που παρέστησαν, που εκφώνησαν τις ομιλίες τους για τη μέρη που έδειξαν και τη δέσμευσή τους να στηρίξουν αυτή την πολιτική. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συνάντησή μας, το οποίο θα αναλάβει να διευθύνει ο Τζάκι Ντέιβις. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Χούμπνερ και να ευχαριστήσω και τους πρώτους μας ομιλητές που μας έδωσαν τέτοια έμπνευση. με Τζάκι Ντέιβις και θα διευθύνω το επόμενο μέρος της συζήτησης. Στόχος μου είναι μιας και μιλήσαμε για το τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε περιφέρειες και πόλεις στο μέλλον της πολιτικής συνοχής, σε αυτό να επικεντρωθούμε για το πώς θα διαμορφωθεί ο ρόλος αυτός όσο προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Θέλω λοιπόν εδώ να συμμετάσχετε όσο το δυνατόν περισσότεροι στην όλη συζήτηση και θα επικεντρωθούμε σε τρία βασικά θέματα όλα κάτω από την, ε, το γενικότερο θέμα της επένδυσης στο μέλλον της Ευρώπης. Την ολοκληρωμένη ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη για τις πόλεις. Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε για τη στρατηγική της, ε, της Ευρώπης για το 2020 και την πολιτική της συνοχής, για την καλύτερη υλοποίηση δηλαδή περισσότερες επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη και τη σημασία της γεωγραφικής διάστασης. Μας το είπε και ο Υπουργό μόλις τώρα. Είναι πολύ σημαντική η γεωγραφική προσέγγιση για να καταφορήσουμε τις σωστές στρατηγικές. Σε αυτά λοιπόν θα επικεντρωθούμε. Αλλά ε, πρέπει να πούμε ότι είναι ζωτική σημασία η περίοδο αυτή για την πολιτική συνοχή. Ήδη ε, υιοθετήθηκε ένα πακέτο μέτρων την περασμένη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριο Χαν να μα παρουσιάσει τα βασικά σημεία για την πρόταση αυτή, ώστε να περάσουμε μετά στι λεπτομέρειε με το πάνελ των ομιλητών μα. Επίτροπε Χαν. Um, Ευχαριστώ, Τζάκη. Αγαπητοί πρόεδροι, πρόεδροι, υπουργέ, ευρωβουλευτές, ε, εκπρόσωποι το, της Επιτροπής των Περιφερειών, φίλοι των Περιφερειών και των Πόλεων. Όπως πάντα είναι ιδιαίτερη χαρά να είμαι μαζί σας και να συμμεριστώ και να συμμερίζομαι μαζί σας κάποια από τα πολύ σημαντικά σημεία και στοιχεία που θα έπρεπε να συζητήσουμε τις επόμενες αυτές κοινέ ημέρες μας. Και αυτές οι ανοιχτές ημέρες, οι μερίδες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, μια συμβολική ανάγλυφη ευκαιρία που δίνει ε, αντανακλά τον ρόλο της περιφερειακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης των πόλεων. Ε, φέτος οι ανοιχτές αυτές οι μέρες ε, διεξάγονται όπως αρκετές φορές προαναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα στρατηγική σημασίας συγκυρία υιοθέτησε το πλαίσιο για τη στρατηγική για την ε, ε, συνοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014 στο 2020 ως Επίτροπος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Χαίρομαι πολύ για τις προτάσεις που έχουν τεθεί επί τραπέζης και με την ομάδα μου και εγώ έχουμε σχεδιάσει αυτές τις προτάσεις και ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις ευρύτερες διαβουλεύσεις που κάναμε από τη δημοσίευση της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή για μας λοιπόν κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε η αποστολή μας ολοκληρώθηκε. Προτού σας παρουσιάσω τα νέα στοιχεία για την πολιτική συνοχή, θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Λειτουργεί η πολιτική συνοχή και συνεισφέρει με αξιόλογο τρόπο για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Έχουμε τεκμήρια που το αποδεικνύουν αυτό από το 2000 στο 2006 1,4 ε, εκατομμύρια θέσεις ε, εργασίας δημιουργήθηκαν μέσω από την πολιτική συνοχή 38.000 για την έρευνα. Επίσης ε, έχουμε και την αντικατάσταση του πακέτου που είχε συμφωνηθεί και αρκετές αλλαγές έγιναν στην Ευρώπη. Ζούμε μια μεγάλη κρίση οικονομική και χρηματοοικονομική. Όλο και μεγαλύτερη πίεση υπάρχει στα δημοσιονομικά και στα οικονομικά, αλλά επίσης και όσον αφορά και τη διάθεση στην Ευρώπη υπάρχει ευρωσκεπτικισμός και απογοήτευση από την άλλη πλευρά οι Ευρωπαίοι ηγέτες επομίστηκαν τις ευθύνες τους και ανέλαβαν νέα μείζωνα πρωτοβουλία για να προαχθεί μια πολύ πιο ανταγωνιστική αηφόρα πολιτική για την ανάπτυξη. Κάνω λόγο φυσικά για την πολιτική της στρατηγικής του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφές ως προς αυτά ότι όχι μόνο πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο της στρατηγικής μας αυτή την πολιτική συνοχή, αλλά πρέπει να ενδυναμώσουμε αυτή την πολιτική καθιστώντας την καλύτερη, ευφιέστερη, πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό εισαγάγαμε νέα στοιχεία στην πρότασή μας για την πολιτική συνοχή μετά το 2013. Θέλουμε η πολιτική συνοχή να γίνει η κύρια στρατηγική για τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κύριο κεντρικό εργαλείο ως μέσο που θα δώσει τη δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να είναι μια πολιτική για όλες τις περιφέρειες και θα δημιουργήσει τη δυνατότητα για επενδύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν θέσεις ανάπτυξης, θέσεις ε, εργασίας. Θέλουμε να μπορέσει αυτή η νέα πολιτική συνοχής να αποδώσει και να είναι το δυνατόν αποτελεσματικότερη. Πώς θέλουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Πρώτον, δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν περισσότερο σε λίγες αλλά κεντρικές προτεραιότητες όπως και αγραφούνται στην στρατηγική μας για την Ευρώπη του 2020. Έχουμε λοιπόν έτσι επικέντρωση σε άξονες. Θα δώσουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις αυτές για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν την μέγιστη επίπτωση και την μέγιστη πρόσθετη αξία. Ταυτόχρονα πιστεύω στεναρά ότι οι προτάσεις αυτές είναι επαρκώς ελαστικές και ευλίγιστες ώστε να δίνουν τη δυνατότητα οι περιφέρειες να μπορούν να επιλέξουν την πολιτική τους για τις επενδύσεις που θα βασίζεται στις δικές τους αναπτυξιακές ανάγκες. Το είπα επανειλημμένα στο παρελθόν. Επικέντρωση, εστιασμός και ελαστικότητα. Στην επικέντρωση όσον αφορά του στόχους του, της στρατηγικής 2020, 11 προτεραιότητες και ελαστικότητα να προσαρμόζονται αυτές οι στρατηγικές στις τοπικές ανάγκες. Αυτά δεν είναι απόλυτα καινούργια θέματα. Έτσι η επικέντρωση και η προτεραιοποίηση θα είναι οι κυριότερες πτυχές στην εταιρική σχέση που προτείνουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών για τις περιφέρειες. Δεύτερον, θέλουμε τα προγράμματα να είναι πιο αποτελεσματικά και για να το καταφέρουμε αυτό προτείνουμε τρία μείζωνα νέα προγράμματα ή τρεις μείζονες πτυχές. Πρώτον, μεγάλη στοχοθέτηση και παρακολούθηση. Δεύτερον, όροι και προϋποθέσεις. Τρίτον, εξπόστο προϋποθέσεις και όροι και αξιολόγηση. Παίρνοντας αυτά τα τρία στοιχεία κλειδιά ένα προς ένα, ποια είναι. Αναπτύσσοντας τι τις επενδύσεις ε, για τα προγράμματα θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχει υπάρξει σωστή προεργασία για αποτελεσματικές επενδύσεις και σαφείς ορισμοί για τη στοχοθέτηση και την επίτευξη αποτελεσμάτων, ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε και να τα αξιολογήσουμε σε ένα διαφανέστερο πλαίσιο για την επιτυχία των πολιτικών αυτών. Θέτουμε το επίκεντρο στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Θα κάνουμε το δυνατόν περισσότερα μετά το 2013 και θα επενδύσουμε τους αναγκαίους πόρους σε ένα ευρύτερο μηχανισμό που θα είναι βιώσιμος και διαφανής. Αυτό σημαίνει ότι οι περιφέρειες και οι χώρες θα πρέπει να ταυτοποιήσουν δείκτες από έναν καθορισμένο κατάλογο δικτών όσον αφορά τη στρατηγική του 2020. Για την αξιολόγηση αυτών των στόχων η αξιολόγηση και η παρακολούθηση είναι κύρια ε, δραστηριότητα θα δούμε αν οι επενδύσεις ε, γίνονται εκεί που οι προϋποθέσεις ε, είναι δεδομένες και επαρκούν. Πολλοί από εσά ε, άκουσαν ήδη τα σχετικά με όρους και προϋποθέσεις, conditionalities. Θα θέλαμε να διατίθενται κονδύλια εκεί όπου υπάρχει αποτελεσματικότητα των όρων, εκεί όπου δεν θα υπονομεύεται τίποτα από όλα αυτά, από, άγνωστο, από άγνωστα στοιχεία. Θα υπάρχει λοιπόν ένας κατάλογος γενικών όρων και προϋποθέσεων που πολύ προσεκτικά θα ελέγχουμε προτού εγκριθεί οποιαδήποτε νέα δράση για την υλοποίηση αυτών των στόχων τα στοιχεία θα είναι δεδομένα, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στον καθορισμό του αν επιτεύχθηκαν ή όχι. Για να το καταδείξω αυτό ανάγλυφα, να αναφέρω την ύπαρξη, για παράδειγμα, της ε, εθνικής και περιφερειακής ε, έρευνας για τις στρατηγικές αυτές, την ύπαρξη δράσεων για την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την επιτυχία στην αποδοτικότητα της εκμετάλλευσης ενέργειας, μείωση εκπομπών ρήπων, υιοθέτηση στρατηγικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τους υδάτινους πόρους, για ένα πρόγραμμα για τις μεταφορές που θα είναι βιώσιμο για την ε, ε, αγορά εργασίας Και, τα και, τα και ούτω καθεξής εφόσον οι προτάσεις αυτές θα ε, εμπεριέχουν σαφείς ενδείξεις για να αμείβονται και να ανταμείβονται τα προγράμματα που θα έχουν τις καλύτερες επενδύσεις. Εδώ δεν έχουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ προγραμμάτων μεταξύ τους. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ευθυγραμμίζονται και θα συμμορφώνονται με τη στοχοθέτηση τα προγράμματα. 5% των κονδυλίων θα διατηρούνται ως απόθεμα απόδοσης ή επίδοσης ώστε μετά από μια ευρία αναθεώρηση να μπορούν να, να απελευθερωθούν. Όλα αυτά σαφώς ε, ε, εμπεριέχονται στο ρυθμιστικό πακέτο που έχει τεθεί τώρα υπό διαβούλευση και συζήτηση. Θα στραφώ τώρα στο θέμα το οποίο πολύ συχνά έχει αναφερθεί κατά τις διαβουλεύσεις ε, <clears throat> μετά τη δημοσίευση της έκθεσης για τη συνοχή Κάτι που ακούγεται εύκολο αλλά που είναι πολύ δύσκολο στην επίτευξή του. Απλούστευση, γραφειοκρατική απλούστευση εξέτασε τρόπους και μέσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η απλούστευση. Θέλουμε να το καταστήσουμε ευκολότερο για τους αποδέκτες και εκείνους που θα υποφελούνται από τα κονδύλια να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια. Αυτό αφορά ενιαίους κανόνες και εναρμονισμένους κανόνες. Όχι μόνο σε σχέση με τα διαφορετικά διαθωτικά ταμεία, αλλά και για την ανάπτυξη της υπαίθρου και για την αυτιλιακή πολιτική και για την αλλιευτική πολιτική. Προτείναμε ένα εύρος κανονισμού που θα έχει κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία για τα πέντε ταμεία. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου και το Ευρωπαϊκό Ναυτιλιακό Ταμείο και το Ταμείο Αλληλείας. Αυτό είναι ένα θαραλέο μεγάλο βήμα για ένα ευρύτερο πλαίσιο συντονισμού και απλούστευσης. Περαιτέρω απλούστευση βρίσκεται επίσης και στην καθημερινή διαχείριση των ταμείων. Οι κανόνες επιλεξιμότητας έχουν εναρμονιστεί μεταξύ των ταμείων. Η απλούστευση του κόστους έχει διευρυνθεί και έχουμε εισαγάγει την έννοια του ετήσιου ε, που θα δίνει την δυνατότητα όσον αφορά ελέγχους ε, να διεξάγονται ετήσια και να δίνουν το πράσινο φως. Για περιφερειακά προγράμματα έχουμε ξεχωριστές ρυθμίσεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη τις εγγενείς, ε, τον εγγενή σύνθετο χαρακτήρα των προγραμμάτων αυτών. Και εδώ πάλι οι κανόνες επιλεξιμότητας έχουν εναρμονιστεί περαιτέρω και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα έχουν περιοριστεί. Επίσης με χαρά μπορώ να ανακοινώσω ότι η έννοια της περιφερειακής συνοχής που συγκεκριμένα αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας έχει τύχει πλήρους προσοχής από πλευράς μας. Οι κανονισμοί οι κανόνες αναφέρονται ρητά σε αυτές τις πτυχές στις πιο απομακρυσμένες περιοχές με την διασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων Ακούσαμε την κλήση, την έκκληση των πιο απομακρυσμένων περιοχών να δοθεί δυνατότητα συνεργασίας με τους γείτονές τους. Εν όπως συνεχίζουμε να ε, επενδύουμε στην αηφόρο ανάπτυξη των ε, αστικών κέντρων τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ συνολικά θα πρέπει από το εθνικό επίπεδο να προκαθορίζονται για ολοκληρωμένες δράσεις στα αστικά κέντρα και στις πόλεις μας. Να ολοκληρώσω. Αυτός ο κατάλογος είναι ο κατάλογος των νέων στοιχείων που αφορά εσάς και αποτελεί ένα κοινό εγχείρημα για όλους μας ο κοινό στόχο είναι η ενίσχυση τη εταιρική σχέση μα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπλοκή των εταίρων στον σχεδιασμό και τη διαχείριση και τη λειτουργία των προγραμμάτων. Οι προτάσει μα θα δίνουν καλύτερε ευκαιρίε για τι περιφέρειε, τα αστικά κέντρα και τι πόλει και τι τοπικέ αρχέ και κοινωνίε να διαδραματίζουν ένα ενεργό ρόλο έχουμε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να προετοιμαστεί η επόμενη γενεά των πολιτικών των προγραμμάτων συνοχής θέτοντας στόχους ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί πρόοδος για να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες της στρατηγική του 2020. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε ότι για την εταιρική σχέση και για κάθε λειτουργικό πρόγραμμα τα κράτη-μέλη θα διοργανώνουν εταιρικέ σχέσεις με τις αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές και άλλες ε, ε, αρχές οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και άλλους τομείς και σώματα που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, την κοινωνία ευρύτερα στην υλοποίηση. Για να μπορέσουν όλα αυτά να προαχθούν θα υιοθετήσουμε και θα προαγάγουμε έναν ευρωπαϊκό διοντολογικό κώδικα προτείνοντας αυτές τη ρύθμιση των εταιρικών σχέσεων για την υποστήριξη αυτών των διεργασιών και για να υπάρξει ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών, εμπειρίας, πείρα και των πρακτικών. Και τέλο, εν κατακλείδη, για την παρουσίαση αυτού του πακέτου δεν μπορώ να ολοκληρώσω χωρίς να στραφώ στο θέμα των δημοσιονομικών πόρων. Τον Ιούνιο έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις για τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια από το 2013 στο 2020. 276 εκατομμύρια ευρώ δίνονται στην πολιτική συνοχή και τα μέσα της και τη νέα διευκόλυνση, την ευρωπαϊκή διευκόλυνση. Ένα τρίτο του προπολογισμού της Ένωσης ε, είναι αυτό. Αυτό είναι σαφές. Δεν ζητάμε περισσότερα χρώματα, ε, χρήματα. Συγγνώμη. Υπό τη σημερινή δημοσιονομική και οικονομική κρίση πρέπει να μπορέσουμε με τους παρόντες διαθέσιμους πόρους να είμαστε πιο ευφυείς και αποτελεσματικοί. Να έχουμε μια πολιτική που θα είναι και πιο φιλόδοξη αλλά και πιο αποτελεσματική. Με ισχυρή συνιστόσα διακυβέρνησης, αποτελεσματικής διαχείρισης μείωσης του γραφειοκρατικού βάρους και αποτελεσματικότητας ε, για όσους εμπλέκονται. Σας έδωσα μια σφαιρική εικόνα του δικού μας οράματος, οράματος για την πολιτική συνοχή. Τώρα εξαρτάται από εσάς, ε, τους ε, Ευρωπαίους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και μέσων, να συνεισφέρετε επικοδομητικά στη συζήτηση τους επόμενους μήνες. Και γι' αυτό θα ήθελα να δραχθώ αυτής της ευκαιρίας και να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία, ιδιαίτερα την Εσβιέτα Μπιενκόφσκα για την σοβαρή εμπλοκή και προσπάθειές τη τους τελευταίους μήνες και τους επόμενους μήνες που έχουμε μπροστά μας. Προσβλέπω λοιπόν και αδειμονώ να ακούσω και να παρακολουθήσω την ανταλλαγή απόψεων που θα ακολουθήσει και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε παθέων, κύριε Πέτροπε. Πολύ σαφή η παρουσία σα και ιδιαίτερα λεπτομερή για τον χρόνο που είχατε στη διάθεσή σα. Ε, όμως θα ήθελα να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα τα στοιχεία που μα ανέφεραν οι μιλητέ μα. Θα χωρίσουμε λοιπόν τη συζήτηση σε τρία τμήματα. Ε, στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, καλύτερη υλοποίηση και γεωγραφική προσέγγιση. Για την κάθε περίπτωση θα δούμε ένα μικρό βιντεοκλειπάκι που θα μα εισαγάγει το κάθε θέμα και ε, θα ξεκινήσουμε με το συγκεκριμένο παράδειγμα του πώ ε, δημορφώθηκαν οι καθημερινέ ζωέ των ανθρώπων από τον αντίκτυπο τη περιφερειακή πολιτική και πώ ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα των διορθωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχή οι πολίτε σε καθημερινό επίπεδο. Για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και μετά την δημοσίευση της Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα είδα ότι υπάρχουν αμέτρητοι ομιλητές στην αίθουσα που θα θέλουν να ζητήσουν το λόγο. Προσπαθήσουμε λοιπόν να καλύψουμε όλου του ομιλητέ, αλλά δίνοντα το δύο λεπτά μόνο στον καθένα στο να προλάβουμε. Θέλω να έχουμε στο δυνατόν πιο πλούσια συζήτηση με όλους ε, εδώ. Και θα προσπαθήσουμε να κλείνουμε το κάθε κεφάλαιο πριν περάσουμε στο επόμενο με όλους τους ομιλητές. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει μετάδοση στο ίντερνετ live και υπάρχει και διαρκή ενημέρωση στο Twitter, στο Europe Regional και επίσης και στο ανάλογο site της Ευρώπης ανοιχτές ημέρες. Υπάρχει όμως και το δίκτυο της Ευρώπης 2020. Η συζήτησή μας όμως δεν θα είναι εικονική, θα είναι με σάρκα και οστά. Θα περάσουμε λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα και θα στραφώ με ένα συγκεκριμένο ερώτημα στην Υπουργό πρώτα. Πριν από δύο χρόνια περίπου, οι πολίτες προέβλεπαν το τέλος της πολιτικής συνοχής όπως την ξέρουμε σήμερα. Όμω ο πρόεδρο Μπαρόζο μα περιέγραψε κάτι που μοιάζει με μια πολιτική τη οποία οι αξίε, και τα ωφέλη είναι ακριβώ τα ίδια. Μια πολιτική για όλε τι περιφέρειες. Γιατί πιστεύετε ότι άλλαξε η προσέγγισή μα. Και γιατί εσεί και όσοι κάθονται στο τραπέζι του Συμβουλίου έχουν τέτοια εμπιστοσύνη στι προτάσει τη Επιτροπή, θα γίνει αποδεκτή μάλλον ή όχι, το πιστεύετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ο λόγος είναι ότι εμείς βρισκόμαστε σε μια πολύ ξεχωριστή συγκυρία χρονικά όπως αναφέρθηκε, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούν μια περίοδο σοβαρής κρίσης. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια πολιτική που θα μπορούσε να μπορέσει να προσαρμοστεί ήπια και να μπορέσει να μεταμορφωθεί σε μια πολιτική για την ανάπτυξη και την πρόοδο της ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση αυτή διεξάγεται και γίνεται επί ολόκληρα τεσσέρα χρόνια και μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι αν υπάρχει μια πολιτική, αν υπήρχε μια πολιτική που θα μπορούσε να μεταφράσει τους στόχους και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για, την, για το 2020 υπό τους όρους καθημερινής ε, πρακτικής ζωής, ε, το μόνο που θα μπορούσε να αναφέρεται σε, στην αποτελεσματική εφαρμογή, η μόνη πολιτική που έχουμε είναι η πολιτική που αποκαλούμε αυτή τη στιγμή πολιτική συνοχής. Πολωνία είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα πόσο αυτή η πολιτική συνοχή μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά αποτελεσματικά. Η, τα ωφέλη αυτής της πολιτικής δεν περιορίζονται σε κάποια χώρα ως αποδέκτη είναι ευρύτερα τα θετικά αποτελέσματα υπέρ όλων και τα στοιχεία αυτά δείχνουν το ότι η πολιτική συνοχή στην Πολωνία έχει θετικότατες επιπτώσεις και σε άλλες χώρες. Σε εμά ειδικά για την Γερμανία, Γαλλία. Ναι, ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Αυτοί είναι οι συντελεστές και οι παράγοντες που βρίσκονται πίσω από την ανάγκη του να συνεχίσουμε να θέτουμε το κέντρο βάρους σε αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ. Έχετε πολύ σπουδαίο έργο μπροστά σα και βεβαίω πρέπει να φύγετε. Α ε, χαιρετήσουμε λοιπόν κυρίε και κύριοι την Υπουργό πριν ε, αποχωρήσει. Σα ευχαριστούμε. Επίτροπε, αν μπορούσα να στραφώ σε εσά να ρωτήσω ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν αγωνιστήκατε ιδιαίτερω για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Εσεί γιατί πιστεύετε, τουλάχιστον είπατε ότι Υπάρχουν περισσότερες, ε, ε, περισσότερες τροφή προς τις επενδύσεις. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια έχουν γίνει επαναστατικές προσπάθειες αλλά και κάπως εντηρητικές ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό. Πραγματικά δεν είχαμε και πολύ χρόνο διότι μια διετία ίσως να ήταν, ίσως και λιγότερο. Όμως προσπαθήσαμε να χτίσουμε αυτά που είχε ξεκινήσει η κυρία Χούμπνερ ως Επίτροπος ε, επί της δικής της θητείας. Εντοπίσαμε συγκεκριμένα κονδύλια, τα στοχεύσαμε και αυτό διευκόλυνε ιδιαίτερα το να μετατοπιστούμε ε, σε μια νέα πορεία. Μπορέσαμε λοιπόν να βασιστούμε στο παρελθόν. Εντοπισμό των κονδυλίων, ε, ευθυγράμμιση όμως. Το σημαντικότερο πιστεύω είναι να πούμε ότι σαφώς Πιστεύουμε πλέον ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να γίνει ε, ε, αντιληπτή και ως επενδυτική πολιτική. Επενδύουμε στους πολίτες και τις περιφέρειες και παίρνουμε πίσω μεγαλύτερο κέρδος από αυτά που αρχικά επενδύσαμε. Γι' αυτό επενδύσαμε με τη θέσπιση τόσων μέτρων. Γι' αυτό συνδυάσαμε την επικέντρωση με την ευελιξία, την ε, παροχή κινήτρων, την τα θέσπιση όρων. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει διάθεση, δομή μάλλον, εταιρική σχέση στην όλη συνεργασία μας. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά εξελίσσεται αυτή η πολιτική και εξελίσσεται κατά τρόπο άριστο για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά μιλάμε για ακραία εξέλιξη. Κυρία Χέμπνερ, όπω είπε ο Επιτροπός, εσείς ξεκινήσατε αυτήν την κοινοτόμο προσπάθεια. Πώς αισθάνεστε για το αποτέλεσμα. Ιδίω επειδή διατηρείται αυτή η αρχή. Μια πολιτική για όλες τις περιφέρειες όλης της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι θα επιβιώσει αυτή η φιλοσοφία μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι οι, πιο, οι μεταξύ μας θα θυμούνται ότι έγινε πραγματική μάχη για να διατηρηθεί η πολιτική συνοχή σε αυτή για τις, όλες τις περιφερειές της Ευρώπης. Τότε ο στόχος 2 ήταν πραγματικά σε σύμπνοια με όσα έλεγαν κάποια κράτη-μέλη, όμως το θέμα είναι να σκεφτούμε και τη φιλοσοφία πίσω από όλα αυτά. Εάν γίνει μια πολιτική για τους φτωχότερους της Ένωσης είναι σαν πολιτική ελιομοσύνης, τότε χάνει και το κύρος της, την προστιθέμενη την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα γινόταν μια πολιτική για την οποία δεν θα καμαρώναμε. Πρέπει λοιπόν να το θυμόμαστε αυτό για πάντα. Δεν πρέπει να γίνουμε μάχη μόνο κάθε πέτεια για τις φτωχές περιοχές. Όχι. Είναι μια πολιτική τόσο πολύτιμη ακριβώ γιατί μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς και να λειτουργήσουν ως κινητήριες δυνάμεις κάποιες περιοχές, περιφέρειες που ήδη έχουν το δυναμισμό τη δυνατότητα να σύρουν πίσω τους και τα υπόλοιπα βαγόνια. Έτσι θα επενδύσουμε στις φτωχότερες περιοχές για να αναβαθμιστούν, να πάνε με όλη την αναξοστοιχεία στον ίδιο ρυθμό και ταχύτητα. Αυτό θέλουμε να γίνει για όλες τις περιφέρειες και είμαι περήφανη διότι πάμε στην κατεύθυνση την οποία χαράξαμε από το 2006 Αποδεικνύει αυτό ότι η πολιτική μας πραγματικά κινητοποιεί τη δυνατότητα ανάπτυξης, τη δυνατότητα εξέλιξης της κάθε περιοχής και κάθε περιφέρειας. Μπορούν να ενδυναμωθούν έτσι οι περιφέρειες σε ένα διεθνοποιημένο πλαίσιο. Και να σας πω ότι κι εσείς υπήρχε μια εξαίρεση πέραν μια εξαίρεση μάλλον, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και εσεί δείχνετε ιδιαίτερη περήφανη. Αλλά ε, σα εκπλήσει το που έχουμε φτάσει σήμερα, κυρία Μπρέσο. Όχι, δεν εκπλήσωμαι. Κάναμε νομίζω πολύ καλή δουλειά όλοι μαζί και με τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών. Το αποτέλεσμα καλώς ήταν αυτό που είναι για τις ε, μεταβατικές λόγου χάρη περιοχές, την νέα αυτή κατηγορία. Αυτό είναι θετικότατο στοιχείο για πολλές από τις περιοχές μας και θα συμφωνήσω απολύτως ότι χρειαζόμαστε ισχυρότερη επενδυτική πολιτική. Ξεκινήσαμε λοιπόν καλά αλλά ας φροντίσουμε να ολοκληρώσουμε και καλά, εφόσον έχουμε ένα τόσο καλό πρόγραμμα στα χέρια μας. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε στο πρώτο από τα συγκεκριμένα μας θέματα. Το έχουμε ήδη θίξει. Τι επενδυτικέ πολιτικέ και τι πολιτικέ συνοχέ τι έχουμε ήδη συζητήσει, αλλά θα επικεντρωθούμε στα στρατηγική του 2020 και την πολιτική τη συνοχή. Λοιπόν, τι μπορούμε να μάθουμε ε, βλέποντα το πρώτο βίντεο ήδη. Ένα παράδειγμα από το πώ ωφελείται κανεί από την πολιτική συνοχή στην πράξη. Εάν έχουμε το κλειπάκι. Λέγομαι Βιμ Κούπερ, είμαι 68 χρονών, είμαι παντρεμένος με τη Μέρη και εδώ και κάποιους μήνες λάβαμε ένα γράμμα για ένα έξυπνο πρόγραμμα. Υπογράψαμε και αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον μετρητή που μας, προτάθηκε για να δούμε πόση ενέργεια καταναλώνουμε εγώ και η γυναίκα μου. Όμω, μάθαμε το εξή, ότι το πλυντήριό μα και το στεγνοτήριο είναι αυτά που καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια. Μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά, να παρουσιάζονται σε μια οθόνη. Επίση, προσέξαμε ότι και για, την, ε, για το πότισμα είναι πάρα πολύ η κατανάλωση. Είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί αυτό το σχέδιο Είμαστε πάρα πολύ θετικοί γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Είναι πολύ καλό που στηρίζετε αυτό το πρόγραμμα. Εγώ συμφωνώ. Uh, Καλώς. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στην πράξη. Ενεργειακή απόδοση και ανανόσιμες πηγές ενέργειας πώς έχει χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση για να το πετύχουμε αυτό. Θα ζητήσω λοιπόν να πάρουν το λόγο όσοι τον έχουν ζητήσει από την αρχή με σύντομες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις προς το πάνελ και μετά θα επανέλθω στο πάνελ και θα τους ζητήσω να απαντήσει. Πρώτον, ο Χαμόν Λουίς Βαρκαθέλ Τσίζο που είναι πρόεδρος της αυτόνομης ε, περιφέρειας της ε, Μούστια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντέβης, κυρία Χιούμπνερ, κυρία Μπρέσο, κύριε Επίτροπε Χάν. Νομίζω ότι οι διάφορες αυτές ε, ανοιχτές ημερίδες που οργανώνουμε δείχνουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία πολύ ενδιαφέρουσα για τους Ευρωπαίους, τόσο για τις πόλεις όσο και για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και κυρίως για όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική συνοχής. Επιπλέον, διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή, α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι περιφέρειες συμμεριζόμαστε αυτό που θέλουμε, δηλαδή η πολιτική σε διάφορα επίπεδα. Κάτι πολύ θετικό προκειμένου να εφαρμόσουμε την στρατηγική μας για την Ευρώπη του 2020. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει σε μερικές γλώσσες, δεν περνάει η διερμηνία, σε όλες ναι. Τώρα είναι εντάξει. Α, τώρα είναι εντάξει. Ωραία. Συγγνώμη για τη διακοπή. Συνεχίστε παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι πράγματι διαπιστώνουμε ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν μεγάλη σημασία στο θέμα της στρατηγικής μας για την Ευρώπη του 2020. Όμως νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίζουμε το γεγονός αυτό για να αποφεύγουμε όσο γίνεται περισσότερο να απομακρυνόμαστε από τους βασικούς στόχου της, στόχους της συνθήκης που είναι η προώθηση των κοινωνικών και περιφερειακών στόχων που μερικές φορές προχωράνε από πάνω προς τα κάτω και δεν γίνονται ε, με αυτόν τον τρόπο που λέγαμε πριν, δηλαδή τη διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα. Το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013 λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο προπολογισμό πρέπει να ευθυγραμμίζεται στην Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 και να διασφαλίζει τη συνοχή και τον συντονισμό στην κοινοτική δράση μέσω των κονδυλίων της. Δηλαδή ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα ως μέσον οι επενδύσεις προς τις περιφέρειες. Τελειώνω, τελειώνω κυρία Ντέβις. Έλεγα λοιπόν ότι συνδέοντας άμεσα τη στρατηγική του 2020 και την εθνική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει την πολιτική αυτή ως εφαλτήριο για να εφαρμόσει τους στόχους της για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Ευχαριστούμε. Η επόμενη παρέμβαση είναι από τον Μισελ Ντελεμπά, που είναι δήμαρχος της Δουκέρκης, από την, την Επιτροπή των Περιφερειών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τόσα έχω ακούσει εδώ από τότε που κάθισε εδώ σε αυτό το κάθισμα. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε για την πολιτική συνοχής. Και συμφωνώ και με αυτά που μας είπε ο πρόεδρος Μπαρόσο και με αυτά που είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από δύο εβδομάδες. Περισσότερη Ευρώπη και λιγότερη επανεθνικοποίηση. Όλα αυτά μου φαίνονται πολύ λογικά, πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Όμως πάντα κάπου κολλάει το πράγμα. Και εδώ θέλω διευκρινήσεις. Λυπούμε που το μήνυμα του Πρόεδρου Μπαρόσο αποδυναμώνεται από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να έχει δεχτεί παρά την άποψη της Επιτροπής των Περιφόρειων και παρά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν δεν κάνω λάθος, υπέρ της ιδέας Μέρκελ-Σαρκοζή να βάλουν τη σπάθα του Δαμοκλή πάνω από τις περιφέρειες απειλώντας με άρση και διακοπή των ε, διαρθρωτικών κονδυλίων για τις περιφέρειες των χωρών μελών που δεν τηρούν το σύμφωνο σταθερότητας. Μα πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο μέτρο να ενισχύσει την πολιτική συνοχής. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς αντιφατικό αυτό. Αναγνωρίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αποφύγει την επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής και επικροτώ. Το γεγονός ότι στήριξε τις προτάσεις για τις ενδιάμεσες περιφέρειες, το γεγονός ότι ασχολήθηκε με την περιφερειοποίηση του μηχανισμού, όλα αυτά είναι πολύ καλά. Όμως, γιατί εξαιτίας λένε τη στρατηγικής 2020 το μενού τελικά, το πρόγραμμα δηλαδή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΦΕΝΤΕΡ για ορισμένες ε, περιφέρειες θα μειωθεί σημαντικά. Γιατί οι Βρυξέλλες να θέλουν πάντα να νομίζουν πως γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα από την τοπική αυτοδίκηση για το τι είναι στο συμφέρον της τοπικής αυτοδίκησης υπέρ της συνοχής και της ανάπτυξης, γιατί το ξέρουν καλύτερα αυτοί. Τέλος, Τέλος, μα ε, ρωτήσεις είπατε να κάνουμε. Ε, ορίστε. Αναρωτιέμαι και για την χρησιμότητα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει από την πολιτική συνοχής και από το σχήμα διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα, με τον οποίο συμφωνώ, 50 δις ευρώ υπέρ του προγράμματος Connecting Europe. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη γνώμη μου, μπαίνει στο δρόμο της ε, περιφερειακής, του περιφερειακού μαγειρέματος με έναν τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά θλιβερός για μένα. Τελείωσα, τελείωσα! Λυπάμαι, έχετε δίκιο, φυσικά και έχετε δικαίωμα να ρωτάτε, φυσικά, αλλά πρέπει να έχουν χρόνο και άλλοι να ρωτήσουν και όλοι εδώ να απαντήσουν. Γι' αυτό και είμαι αυστηρή. Έτσι μου ζήτησα να κάνω, αυτό κάνω. Επόμενο... Επόμενη παρέμβαση ο Μάικλ Σάιντερ, ο οποίος είναι δήμαρχος στην Σαξονία και πρόεδρος του τοπικού, ε, της, μάλλον της ομάδας του ΕΛΚ ε, στην Επιτροπή Περιφερειών. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Υπό αυτή την ιδιότητά μου θέλω να πω κάτι ως πρόεδρος της ομάδας του ΕΛΚ. Εξ ονόματος της ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών θα ήθελα στην Επιτροπή και ιδιαίτερα στον Επίτροπο Χάν να δώσω συγχαρητήρια για το πακέτο το οποίο μας παρουσίασαν τους τελευταίους μήνες με το πολιετές πλαίσιο και το πακέτο των σχεδίων κανονισμών. Άνοιξαν την πόρτα προς το μέλλον για την πολιτική συνοχής και οποίο παρακολούθησε τις συζητήσει τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Υπήρχαν πολλοί αντίπαλοι και πολλέ επιφυλάξεις για την πολιτική συνοχή. Με τις προτάσεις σα διασφαλίσατε ότι στο μέλλον η πολιτική συνοχή με νέα στοχοθέτηση θα προχωρήσει. Και προτού ξεκινήσει κανείς να συζητά κάποια πράγματα ή να ασκεί επικρίσεις, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσει θερμά εσάς. Εσείς είσαστε οι πραγματικοί φίλοι των περιφερειών με τις προτάσεις σας, διότι η πολιτική συνοχής πρωτογενώς διεξάγεται φυσικά στις περιφέρειες και το ίδιο και για τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών καλοχαιρετήσαμε αυτή τη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Είπαμε θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να πετύχει. Αναπτύξαμε την ιδέα και προχωρήσαμε με την ιδέα της εταιρικής σχέσης, της δομικής διαφροντικής σχέσης των περιφερειών για αυτή τη στρατηγική. Διαβάζοντας τώρα αυτές τις προτάσεις πρέπει να πω ίσως είμαστε υπερβολικά επιτυχείς με τις ε, ιδέες μας

πρέπει ακριβώς να συζητήσουμε μήπως τώρα η πολιτική συνοχής μονομερός διαμορφώνεται υπό το πρίσμα της πολιτικής για το 2020 και τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Η πολιτική συνοχή είναι κάτι ευρύτερο, έχει μακροπρόθεσμους στόχους, είναι πολυσχηδής και πολυδιάστατη και ε, με ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τις περιφέρειες. Δεν θέλω να δώσω κάποια αξιολόγηση από πλευράς μου, τα θέματα θα τα συζητήσουμε διεξοδικά τους επόμενους μήνες, θα συντάξουμε γνωμοδοτήσεις και με το Κοινοβούλιο επικοδομητικά και με την Επιτροπή θα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Χαιρόμαστε διότι για πρώτη φορά ξέρουμε ότι έχει μέλλον η πολιτική συνοχή πλέον. Σας ευχαριστώ. Υπουργός της Νότιας Αυστρίας για τα θέματα των γυναικών. Ναι, και σε σχέση με την, τον εντοπισμό των προκλήσεων και των κέντρων βάρους όσον αφορά τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και υπό το πρίσμα μας της κάτω Αυστρίας έχουν τεράστια σημασία. Καινοτομία, έρευνα, ανάπτυξη, τεχνολογία ανήκουν σίγουρα στα κεντρικά σημεία ως άξονες μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα κάποιες σκέψεις να σας παρουσιάσω όμως για την ελάχιστη πρικοδότηση για τα κονδύλια για κάθε έναν από αυτούς τους άξονες. Εγώ πιστεύω ότι η ισόρροπη πρικοδότηση και η ισόρροπη συμμετοχή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή είναι αρκετές επιχειρήσεις ε, στις περιφέρειες παρούσες για να μπορέσουν να καλύψουν αυτούς τους τομείς. Δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιες περιφέρειες να έχουν ισχνή παρουσία και να μείνουν πίσω είναι κάπως ασαφής η έννοια της καινοτομίας θα έλεγα. Ωστόσο υπό το δικό μου πρίσμα θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευρύ ορισμό ως ε, ε, γραμμή εκκίνησης και τα προϊόντα και οι διεργασίες ε, ως καινοτομία και τουριστικές καινοτομίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και εδώ πάλι ο στόχος είναι περιφερειακή διαφοροποίηση η Ευρώπη των περιφερειών είναι ετερογενής, ε, ετερόκλητη, δεν είναι ομοιογενής. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να συμπορευθούν και να μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης. Τώρα στοχεύουμε, πορευόμαστε σε μια ξεχωριστή πορεία υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημαντικό όμω είναι να δούμε και τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις που θα μπορούν να ενισχυθούν. Οι μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές δημιουργούν πολλές θέσεις απασχόλησης ε, και πολλές φορές ε, θα πρέπει να δούμε την δυνατότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων να εξοπλίζουν ή να δίνουν τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα εφόδια προς αυτές τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να έχουμε περιθώρια λοιπόν τα οποία θα είναι επαρκή οι όροι και προϋποθέσεις και η χρήση των όρων και προϋποθέσεων αντιμετωπίζουμε με, με κάποια επιφύλαξη αυτό το πεδίο. Σε ένα ομοσπονδιακό κράτος με ομοσπονδιακή δομή όπως ε, στην Αυστρία δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Έχουμε ομοσπονδιακά κρατήρια, κρατήρια και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν όλα αυτά μέσα στο εθνικό πλαίσιο να λειτουργήσουν και πώς θα μπορέσει να υπάρξει λογοδοσία για όλα αυτά. Τελευταίο σημείο τα ε, λειτουργικά μικρά προγράμματα, η λειτουργικότητά τους πρέπει να διασφαλιστεί. Τα μέτρα όχι μόνο να αφορούν τους φορείς των προγραμμάτων, αλλά να υπάρξει απλούστευση. Απλούστευση στο γραφειοκρατικό και διοικητικό τομέα, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστούμε. Ο τελευταίος Χέγγεν, υπουργό Δικαιοσύνη στη Γερμανία, στην περιφέρεια του Τέριεν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε Μπρέσο, αξιότιμε κύριε Χάν. Εκεί, στη μέση, ναι, ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για να εντοπίσουμε που βρίσκεστε. Πώς είπατε, ναι εντάξει τώρα, μπορώ να συνεχίσω. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι μέλος από τα νέα κρατήδια της Ομοσπονδιακής Γερμανίας μετά την ενοποίηση. Θέλω να καλοχαιρετήσω και να ευχαριστήσω προσωπικά για την αλληλεγγύη που εξέφρασε τα τελευταία 20 χρόνια τον Επίτροπο Χάν. Συνολικά στην Θουριγγία πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ είχαμε από τα Ευρωπαϊκά Διαθροτικά Ταμεία από το 1991 που μας δόθηκαν. Ήταν μια καλή επένδυση, αποτελεσματική επένδυση θα έλεγα, προς όφελος συνολικά της κοινωνίας μας και πιστεύω ότι δεδομένη της σημερινή ε, συζήτηση για την, οικονομική μας ε, ε, κρίση και οικονομικά προβλήματα ευχαριστούμε ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή κοινότητα έναντι των νέων κρατηδίων, των νέων χωρών της Γερμανικής Ομοσπονδίας, πρώην Ανατολικής δηλαδή Γερμανίας, για την βοήθεια και αλληλεγγύη. Και επίσης έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να υπάρξει ενδυνάμωση που χρειάζεται σε σχέση με την κρίση. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερα κοινά στοιχεία για όλους και λιγότερες θα έλεγα μονομερείς αποκλίνουσες πορείες όπως το ανέφερε ο Επίτροπος Χάν, να επενδύσουμε στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση, σημαντική ιδέα και συζήτηση αυτή. Η μελλοντική πολιτική συνοχής βρίσκεται έτσι στη σωστή πορεία, στη σωστή κατεύθυνση. Εύχομαι σε, όλους μας, σε μας καλή επιτυχία σε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό εγχείρημα. Uh, Πριν uh, επιστρέψουμε στο πάνελ για να δούμε μήπως υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις σχόλια. Παρακαλώ πείτε ποιος είσαστε, ποιον εκπροσωπείτε και να είσαστε σύντομος. και πείτε που είσαστε για να μπορεί να σας εντοπίσει και η κάμερα, έτσι, γιατί είπαμε ότι περνάμε στο διαδίκτυο, οπότε να μπορούμε να σας εντοπίσουμε. Σάκ Μπλον λέγομαι, Γαλλία, και χαίρομαι που κύριε Επίτροπε, και ξέρω ότι έχετε αγωνιστεί γι' αυτό, για τις διάμεσες ζώνες ή περιφέρειες. Όμως, από την άλλη δεν άκουσα τίποτα για τις ορεινές περιοχές, για τα βουνά. Ενώ στη συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο το οποίο δημιουργεί την εδαφική συνοχή, λέει, σε παρένθεση, ε, τα νησιά και τα βουνά με ειδικέ πιστώσει υπέρ των ορεινών περιοχών για να πετύχει λοιπόν η εδαφική συνοχή. Θα το κάνετε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα φροντίσω να απαντήσει λίγο η Επιτροπή. Διάφοροι ευρωβουλευτές νομίζω είχαν πει ότι ήθελαν να πάρουν το λόγο κάποια στιγμή. Μήπως κάποιος τώρα. Ο κύριος Βάμπακ ή ποιος. Παρακαλώ. Εσεί. εσείς. Κάτεμπαχ, 16 χρόνια στην κοινοτική πολιτική και 10 χρόνια στο κρατήδιό μας ε, με σημαντική ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής και υπό το, την προσωπική μου πείρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο Χάν προσωπικά που στην Περιφερική Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο πάντα με πολύ θετική εταιρική σχέση ερχόταν σε εμά και μας προσφωνούσε και μας ενημέρωνε και για την Επιτροπή Περιφερειών που ακριβώς το θέμα της προαγωγής και υποστήριξης των ε, ε, ενδιάμεσων περιφερειών ως κατηγορία έχουν συνεισφέρει θετικά. Για τις ενδιάμεσες περιφέρειες είναι πολύ σημαντική υπόθεση ώστε να μπορέσουν τα ταμεία στο μέλλον να συνεργαστούν πολύ πιο αποτελεσματικά εκεί που έχω κάποια προβλήματα, όχι μόνο κάποια προβλήματα, αλλά σημαντικά προβλήματα και το είδαμε και με το βιντεάκι, είναι πώς η πολιτική συνοχής επιτόπου θα αντανακλάται και ποιες επιπτώσεις θα έχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν έχω καμία κατανόηση λόγω κακής συμπεριφοράς και στάσης, κακής δραστηριοποίησης στα κράτη-μέλη για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε φταίξιμο που έχουν από πλευράς της ε, πολιτικής τους να την πληρώνουν, να πληρώνουν τα σπασμένα οι περιφερειακές κοινότητες. Και στο ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ μεγάλη κατανόηση πρέπει να δείχνεται περιφερειακά για την κοινωνική συνοχή και την πολιτική συνοχή σε αυτών των περιφερειών. Εδώ δεν πρέπει να υπονομευθεί η αλληλεγγύη. Γι' αυτό το σημείο θα πρέπει να προβληματιστείτε και δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε να υπονομευθούν αυτές οι αρχές. Ευχαριστώ. Παρακαλώ εσείς. Πολύ σα ευχαριστώ. Είμαι μέλο τη Επιτροπή Περιφερειακή ε, ανάπτυξη. Θα ήθελα να πω ότι εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικέ συνοχή είναι ουσιοδέστατε για να βρούμε διέξοδο και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα θεμελιώδη θέματα για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι οι σημαντικέ ασυμμετρίε ανταγωνιστικά που υπάρχουν και οι ασυμμετρίε μεταξύ των περιφερειών μα. Αυτά σε σχέση με μια πολιτική στην συγκυρία που βρίσκονται τα κράτη-μέλη με δυσκολίες για να διασφαλίσουν επενδύσεις και δυσκολίες να προαγάγουν την ανάπτυξη. Και απαιτείται να δούμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες για την χρηματοδότηση των επενδύσεων, για τα διαθροτικά ταμεία που διαδραματίζουν εδώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτούς τους λόγους η δυνατότητα απλούστευσης αυτών των ταμείων και των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης των κονδυλίων τους είναι ουσιοδέστατο στοιχείο ώστε οι χώρες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να μπορούν να έχουν μια δυνατότητα να έχουν 10% είναι πολύ σημαντικό να μην περιοριστούμε σε αυτό το 10% στο εύρος. Να υπάρχουν και οι περιφέρειες που σήμερα θα μπορούν να ε, δραστηριοποιηθούν. Έχουμε το όριο 85%. Πρέπει η επέκταση 10% να ληφθούν υπόψη για όλες ε, τις περιφέρειες και τις ενδιάμεσες περιφέρειες. Επίσης, οι μακροοικονομικοί όροι και προϋποθέσεις. Φαίνεται εδώ να υπάρχει μια αντίφαση και αντίθεση σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Αυτά τα κονδύλια είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτέ τι περιφέρειε. Να συμμετέχουν στι δεσμεύσει που θέσπισαν τα κράτη-μέλη για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Το απλό γεγονός της αυτόματης παρέκκλησης όταν δεν θα υλοποιούνται οι στόχοι είναι μια παραβίαση αυτών των αρχών. Ευχαριστώ. Να πω απλώς και να τονίσω σε αυτή τη φάση ότι έχουμε και το επόμενο κεφάλαιο. Θα μιλήσουμε για την καλύτερη υλοποίηση, τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε θα επικεντρωθούμε στο θέμα των όρων και των προποθέσεων και θα δούμε το εξωτερικό και το εσωτερικό επίπεδο. Θα δούμε και την απλούστευση. Οπότε για την ώρα ας προσπαθήσουμε να παραμείνουμε στο τι γίνεται με την Ευρώπη του 2020 και τη σχετική στρατηγική να, καλύψουμε, να χωρίσουμε λοιπόν τα θέματα σε τρία κεφάλαια. Ο Σον Κέλλη, πού πήγε. Σον Κέλλη, έχετε το λόγο. Μόνο ένας ομιλητής και μετά το πάνελ. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Χαίρομαι που βλέπω εδώ κάποιους υπέροχους ανθρώπους, ιδίως εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών. Νομίζω σωστά υπόθηκε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, αλλά πάνω απ' όλα ισότιμη Ευρώπη και περισσότερη αλλά και πιο ισότιμη. Έτσι λοιπόν, τέτοια αποτελέσματα μπορούμε να τα πετύχουμε με την πολιτική συνοχή. Και είναι επιτυχής η πολιτική συνοχή, ιδίω αν δει κανεί πόσε είναι οι περιφέρειε που συγκλίνουν, έχουν ακολουθήσει του στόχου σύγκληση. Είδαμε τον κύριο με το τσιγκελωτό μουστάκι πόσο ικανοποιημένο ήταν στο κλειπάκι. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμη περισσότερα καλά που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την πολιτική. Ε, και θα πρέπει να τονιστούν τα θετικά. Να δούμε τα ωφέλη του να ανήκει κανείς στην Ευρώπη, ιδίω να δοθεί έμφαση στην πολιτική συνοχή στο μέλλον. Μία από, ένας από τους λόγους της επιτυχίας της πολιτικής συνοχής και ίσως και αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης είναι η ιδέα της δημιουργίας των μεταβατικών περιοχών, κάτι που συζητήθηκε διεξοδικά, διαμακρών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Επίτροπο ίσως, ή τον Επίτροπο, να μας πούν αυτό πώς το διαβλέπει σε σχέση με την ε, στατική το 2020, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι θα γίνει συνολικά ως προς την πολιτική συνοχή. Μάλιστα τώρα να επιτρέψουμε στο πάνελ, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που ετέθησαν, θα ήθελα εάν γίνεται να δούμε ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν στο τέλος. Αλλά το θέμα των όρων και προποθέσεων τέθηκαν ξανά και ξανά. Η Ευρώπη της στρατηγικής του 2020, οι διαφοροποίησεις μεταξύ των περιοχών, η μείωση των επιλέξιμων προγραμμάτων. Πολλά από αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με την επιλεξιμότητα. Προσπαθώντας λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε την πολιτική συνοχή με την Ευρώπη του 2020, τελικά μήπως έχουμε πάει πολύ μακριά, μήπως έχουμε γίνει πολύ αυστηροί ώστε να απαιτούμε από τις ε, διάφορες περιφέρειες να κάνουν αυτό που πρέπει για να πετύχουν κάτι. Θα δώσω σε εσάς το λόγο πρώτα, κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά πολύπλοκο το ερώτημα, όμως οπωσδήποτε έχουμε μια κάποια ανησυχία διότι η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, την οποία και τη συμμεριζόμαστε και εφόσον βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής συνοχής, ίσως τελικά να γίνει ένα κλουβί, ε, να γίνει περιοριστική σε κάποιες δεδομένες ε, περιπτώσεις, ιδίως από την ενταφική την άποψη. Μην ξεχνάμε ότι οι στόχοι της πολιτικής συνοχής είναι πολύ σαφώς καθορισμένοι ε, το να τους ορίζουμε, να τους κάνουμε τόσο λεπτομερή στην περιγραφή γίνεται κάτι σαν ένα χρυσό κλουβί, δηλαδή δυσκολεύουμε τα πράγματα. Θέλουμε να υπάρξει πραγματική συμμετοχή των περιοχών και των περιφερειών στον ορισμό των συμβάσεων. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα προγράμματα των ε, περιφερειών στην στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 αλλά όπως η κάθε επικράτεια ξεχωριστά μπορεί να την ε, προσδιορίσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει η περιφερειακή ανάληψη ευθύνη που προτείνουμε και οι τοπικές συμβάσεις να είναι πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Κυρία Χούμπνερ, βλέπετε και εσείς τις συμβάσεις ως το κλειδί για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ακρίβειας. <clears throat> Κοιτάξτε, κανονικά ευελιξία σημαίνει εξαίρεση από έναν κανόνα. Ε, Κάποιε φορέ οι κανόνε είναι και πολύ περίπλοκοι. Οπότε πάντοτε υπάρχει πρόβλημα, κάποια πρόκληση τέλο πάντων για όσου ε, κοιτάζουν το νομικό πλαίσιο. Την πρόκληση την αντιμετωπίσαμε προ πενταετία και τώρα την αντιμετωπίζουμε προσπαθώντα να βρούμε την ε, σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξία και περιπλοκότητα. Όμω, Γι' αυτό ακριβώς ε, επινοήσαμε αυτή τη στατική προσέγγιση. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία για να διασυνδέσουμε τις ευρωπαϊκές περιοχές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτήν λοιπόν την πρόκληση πρέπει να την ε, αντιμετωπίσουμε βρίσκοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ των στόχων του 2020 και τι εδαφικές ιδιαιτερότητε. Να προσθέσω όμω ακόμη κάτι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μια δικασία μόνο που ξεκινάει από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά και το ανάποδο. Δηλαδή χρειάζονται τοπικές προσπάθειες, ε, οι προσπάθειες των περιφερειών, ώστε να εντοπίσουν τα δυνατότητές τους, τους στόχους τους μέσα από αυτή τη στρατηγική του 2020. Να μπορέσουν λοιπόν να διασυνδεθούν οι ίδιοι με τους ευρωπαϊκούς στόχους με 11 προτεραιότητες που ήδη έχουν προταθεί. Εσείς λοιπόν, εσείς πρέπει να σκεφτείτε και αυτό θα πρέπει να είναι μια αμφίδρομη διαδικασία ώστε να πετύχουμε μια σωστή ισορροπία και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και μέσω των συμβάσεων. Σας ευχαριστώ. Αυτό το ζωτικό ερώτημα της ευελιξίας σε σχέση με την ε, υπερβολική ακρίβεια, τη στόχευση. Τελικά είναι πολύ αυστηρός ο κατάλογος των περιοχών. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες βέβαια ακούσαμε ότι υπάρχει κάποια επιλογή, αλλά και το θέμα των μεταβατικών περιοχών. Υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις γι' αυτό. Μπορείτε να το σχολιάσετε παρακαλώ, Επίτροπε. Τώρα θα μιλήσω για μια διαφορά, μια αλλαγή γερμανικά πάλι. Για το θέμα αυτό μεταβατικών περιφερειών ή ας το πω αντίστροφα ε, για τους στόχους της Ευρώπης 2020. Τα είδαμε τα πράγματα ήδη σήμερα. Σχεδόν πάνω από 90% των κονδυλίων του προϋπολογισμού στην περιφερειακή πολιτική μπορούν να θεωρηθούν υπό την στοχοθέτηση του 2020 και των αξώνων της στρατηγικής του 2020. Δεν επινοούμε τον τροχό εκ νέου καθόλου. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι μέσα στο πλαίσιο αυτών δηλαδή της διασφάλισης της αρχής της ολοκληρωμένης προσέγγισης ως αφετηρία, να υπάρχει θεματολογικά επικέντρωση, εστιασμός στις πτυχές όλου αυτού του φάσματος. Και αν σας πω και όταν σας λέω προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην καινοτομία και μέσα στο πλαίσιο της καινοτόμας δράσης, αυτά μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο πρέπει να ενταχθούν και όχι μόνο να αφορούν τεχνολογική καινοτομία ή το μάρκετινγκ για την παροχή υπηρεσιών με καινοτόμο τρόπο ή διοικητικέ καινοτομίε, όχι μόνο αυτά. Όταν σκεφτόμαστε την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενεργειακή εξοικονόμηση, τότε είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα ως πεδίο δράσης ε, θεματολογικά, ώστε μια ακριβέστερη ανάλυση οδηγεί στο να μην χρειάζεται κανείς να ανησυχήσει ότι με τις προθέσεις του θα, θα βρει προσκόμματα ή εμπόδια. Αυτό που θέλουμε εμείς ε, είναι να υπάρξει επικέντρωση στη σωστή δράση. Δέσμευση για σαφείς στοχοθετημένους και ποσοστοποιημένους στόχους στόχους ώστε να ανταποκρινόμαστε στη στοχοθέτηση της Ευρώπης 2020 ως στρατηγική. Αυτό το μάθημα, αυτή τη στοχοθέτηση πρέπει να έχουμε μάθει από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Πρέπει ευρωπαϊκούς στόχους σε εθνικά και περιφερειακά επίπεδα να αναλύσουμε και να αρθρώσουμε για να είμαστε αποτελεσματικοί και ρεαλιστές. Στη στοχοθέτηση πολλές φορές δεν υπάρχει μια άμεση διασύνδεση. Όταν η Ρουμανία έχει ποσοστό έρευνας κάτω από 1%, η Σουηδία 4%, τότε αυτά τα 3% δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά ούτε για τον μεν ούτε για τον δε. Πρέπει ρεαλιστικούς στόχους να θέσουμε λοιπόν το άθροισμα αυτών των φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών και κοντά στην πραγματικότητα στόχων για τις περιφέρειες θα δώσουν αυτό το 3%. Για τις ε, ενδιάμεσες περιφέρειες αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι μέσω μιας αναδιαμόρφωσης ε, της ε, αρχιτεκτονικής για τη χρηματοδότηση ιδιαίτερα με το σκεπτικό ότι για τη μελλοντική χρηματοδοτική περίοδο ενίσχυσης λιγότερο, πώς να το πω, less developed regions θα έχουμε λιγότερες μη ανεπτυγμένες ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες από ό,τι σήμερα θα, από το 84% θα έχουμε ένα 68% λιγότερο αναπτυγμένων και η ανταλλαγή μεταξύ των λιγότερων αναπτυγμένων και των μεταβατικών περιφερειών θα μας δώσει μια δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί. Ένα επιχείρημα να σας δώσω, ένα αριθμητικό μέγεθος, ένα αριθμό που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί αυτή η μεταβατική κατηγορία περιφερειών για αυτή, την για αυτή τη χρηματοδοτική περίοδο. Δεν είναι κάτι ιστοδιεινεκές ή αιώνιο αυτό που κάνουμε με διαρκή ε, χαρακτηριστικά, αλλά για τις περιφέρειες αυτές ε, με μέσο ΑΕΠ 53% και για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές που έχουν 122% του μέσου εισοδήματος το χάσμα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το 75% που ήταν στόχος. Οι μεταβατικές αυτές περιφέρειες βρίσκονται μέχρι το 85%. Όμως το ποσοστό απασχόλησης, employment rate, είναι σημαντικό στοιχείο που δίνει χαρακτηριστικά πραγματικής απασχόλησης πραγματικά απασχολούμενων σε μια τέτοια περιφέρεια. 63% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, 73% σε πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 10% διαφορά στις ε, μεταβατικές περιφέρειες 67%. Χρειαζόμαστε αυτή την κατηγορία λοιπόν ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτές τις περιφέρειες. Ευχαριστώ. Ωραία, να περάσουμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο θέμα μας, αλλά πρώτου από αυτό να ε, αναφέρω και τα έπαθλα που δίνονται στις διάφορες περιφέρειες. Τα βραβεία από το 2008 το 2013 θα ξεκινήσουν μάλιστα να, απο, να απονέμονται αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής που θα συζητούμε και εμείς. Πολλά από τα βραβεία λοιπόν αυτά, η ευφύ ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη, η ενταξιακή ανάπτυξη, ε, διασυνδέονται και με τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Ε, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα ληφθούν ε, οι πρώτε υποψηφιότητε. Η προθεσμία βρίσκεται στον ιστοτοπό μα σε μόλι τι σχετικέ πληροφορίε. Τώρα, αυτό έχει να κάνει με την επικοινωνία και τι πληροφορίε που διαθέτουμε και γι' αυτό ακριβώ μα απασχολεί και το δεύτερο θέμα μα. Η υλοποίηση, τα αποτελέσματα. Ε, ο Επίτροπος μας είπε ότι θέλει ένα μεγάλο άλμα πρόοδου ώστε να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα και επιδόσεις από την πολιτική συνοχή του ομιλητέ μα. Είδαμε να γίνονται σχόλια για το θέμα αυτό, αλλά πρωτοηγουμένω α δούμε το φιλμάκι μα. Amal, Amalia. Λέγομαι Αμάλ Γιασμίμα από το Κουρδιστάν ε, του Ιράκ και έχω ζήσει στο Κατίνα Χόλμ στη Σουηδία για δύο χρόνια τουλάχιστον. Η ιδέα μου ήταν να αρχίσω τη μικροοικονομική στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να την χρησιμοποιώ και χρειάστηκα βοήθεια και άρχισα να συνεργάζομαι με αυτό. Όταν ε, ξεκινεί, ξεκινά κανείς την επιχείρησή του στη Σουηδία ε, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία. Όμως ε, τα μικρο, μικροοικονομική πίστοση με βοήθησε για να μάθω με το πρόγραμμα αυτό σε ποιον απευθυνθώ, τι να κάνω και όταν ξεκινούσα ε, καλά πήγαιναν τα πράγματα, όμως τώρα το κέρδος μου έχει διπλασιαστεί. Uh, Ωραία. Είδαμε λοιπόν πώ η ΑΜΑΛ μπόρεσε να ξεκινήσει την επιχείρησή τη, αντιμετωπίζοντα κάποιε δυσκολίε τη. Μπορεί λοιπόν μια πολιτική γενικότερα να δώσει τέτοια αποτελέσματα όπω για την ΑΜΑΛ. Πολλοί έχουν ζητήσει πάλι τον λόγο από πριν. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Κούγκα, ο οποίο είναι μέρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μέρο τη ομάδα Άλντε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στην κυρία, μάλλον. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χούμπνερ μα είπε ότι το 2005 υπήρξε ολόκληρη πάλι για να διατηρήσουμε τότε την πολιτική συνοχή. Πράγματι, πολεμήσαμε σκληρά και νομίζω ότι πάλι δεν θα μπορεί να γίνει με κάποια κρατημέλη για να την κρατήσουμε. Λοιπόν, για όσου θέλουν να κρατήσουν την πολιτική συνοχή, θα πρέπει να συσπηρωθούμε, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το πετύχουμε. Ναι, Επίτροπε, έχετε δίκιο. Θα πρέπει να είναι και επενδυτική πολιτική αυτή. Όχι μόνο μια πολιτική δαπανών. Θα πρέπει οι σωστέ επενδύσει να γίνονται ώστε να γίνουν και οι διαφορέ που θέλουμε στι καθημερινέ ζωέ των ανθρώπων. Αυτό θέλουμε να δούμε να συμβαίνει περισσότερο από εμά. Ε, οι περισσότεροι θέλουν και καλύτερε περιοχέ και στι καλύτερε περιοχέ κάτι τέτοιο και στι φτωχότερε. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να είναι ο προσανατολισμό μα, διότι αυτό που κάνουμε δεν είναι να δαπανούμε τα χρήματα για το τίποτα. Όχι. Εάν έχουμε σωστό στοχεύσει, θα πάνε όλα καλά για τα επόμενα δύο χρόνια στο North έχουμε μια, ένα από τα πρώτα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε μεταξύ του 2000 και το 2006. Ένα ειδικό επενδυτικό ταμείο. Επενδύσαμε στι τοπικέ επιχειρήσει και το ταμείο αυτό ακόμη παίρνει κέρδη από τι επενδύσει που αρχικά είχε κάνει και ακόμη αποφέρει κέρδο στι τοπικέ επιχειρήσει. Φανταστείτε και για τα επόμενα χρόνια θα κρατήσει αυτό. Μέσα στην ίδια μα την περιφέρεια επίση διατηρήσαμε, κρατήσαμε το 54.000 δουλειέ θέσεις εργασίας και ένα τρίτο εκατομμυρίου ε, πολιτών μπόρεσε να καλυφθεί ε, από την άποψη της απασχόλησης. Να ποια είναι η διαφορά που μπορεί να μας κάνει η πολιτική συνοχής. Και για κάτι που υπόθηκε σήμερα εδώ πέρα και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Πρέπει τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο να τους εμπλέξουμε γιατί το να μιλάμε τις εθνικές κυβερνήσεις σε τοπικό επίπεδο δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Η εθνική κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη όπως οι ντόπιοι Γι' αυτό λοιπόν το 5% που έχει στοχευθεί ως κονδύλια για τις πόλεις, το εγκρίνουμε. Χρειάζεται αυτή τη στήριξη να τη λάβουν οι πόλεις. Για την ίδια του την αύξηση και την ανάπτυξη, μάλλον και την ανανέωση. Όμως θα πρέπει ε, να εμπλέκονται οι τοπικοί παράγοντες και στο σχεδίσμα των προγραμμάτων. Ιδάλλως θα υπάρξει αποτυχία. Χρειάζεται λοιπόν μια αμφίδρομη διαδικασία και από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω και για τις διάφορες προϋποθέσεις και όρους. Καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο αυστηρές πλέον οι προϋποθέσεις, όμως καταλαβαίνω ότι αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν. Υπήρχε ένα σύνολο όρων, το 5% της επίδοσης που έπρεπε να αποδοθεί σε όσες περιφέρειες πετύχαιναν τους στόχους που είχαν ε, θέσει οι ίδιοι του εαυτούς τους. Τότε έπαιρναν την επιδότηση. Εδώ λοιπόν είχαμε τη μέθοδο του καρότου και του μπαστούνιου αλλά εδώ τότε μάλλον είχαμε το καρότο και τον μπαστούνι, τώρα έχουμε μόνο το ένα. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ένα κώδικα καλών πρακτικών από τι ίδιε τι περιφέρειες για να αποφύγουμε τα περισσότερα προβλήματα. Πώ θα γίνει τώρα όλο αυτό, Επίτροπε, δεν ξέρω. Καταλαβαίνω από τι συζητήσει που έχουν γίνει με επισήμου ότι ακόμη δεν είναι σαφέ τι μηχανισμό θα προβλεφθεί για να μπορέσουν οι περιφερειακέ πόλει να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Τα εθνικά προγράμματα ήδη έχουν ε, σχεδιαστεί, όμως δεν αρκούν. Θα πρέπει να μας πείτε πώς τα προγράμματα στο εθνικό επίπεδο θα εμπλέξουν τις τοπικές ε, αρχές και τις περιφερειακές για να μπορέσουν να διατεθούν τα κονδύλια. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ζαϊκάτα, ε, δήμαρχος της Πολωνίας. Θα, καλύτερα να πείτε μόνοι σας το όνομά σας, γιατί φαντάζομαι ότι το έγδαρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προφορά του ονόματός μου ήταν η καλύτερη που έχω ακούσει στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου πρώτα να αναφερθώ σύντομα σε κάποιες ουσιώδεις αρχές, βασικές αρχές η πολιτική συνοχή σχεδιάστηκε για να μειωθεί το χάσμα όσον αφορά την ανάπτυξη διαφορετικών κρατών μελών και διαφορετικών περιφερειών. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σε μία και ίδια περιφέρεια υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές διαφορές και υπάρχουν λόγοι να έχουμε την εκτίμηση και δράση για να μειωθούν οι διαφορές που υπάρχουν ακόμα και σε μία και ίδια περιφέρεια. Έχουμε στην περιφέρειά μας ε, δραστήριες ε, πόλεις ε, και αστικά κέντρα και αρκετά κοντά έχουμε ζώνες πολύ χαμηλότερου ποσοστού ή επίπεδου ανάπτυξης. Αυτή ακριβώς η πτυχή της πολιτικής συνοχής δεν θα πρέπει να αγνοηθεί, να, δεν πρέπει να παραμεληθεί στις σκέψεις και στον προβληματισμό μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Στις περισσότερες πολωνικές περιφέρειες, στις πιο πολλές, οι πιο πολλές ε, τα πήγαν καλά. Η πολιτική συνοχή είχε εποφε... Ε, ε, ωφέλησε αυτές τις περιφέρειες και έχουμε και μεταβατικής κατηγορίας περιφέρειες, όμως πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Και Γυρνώντας στην αρχή της παρέμβασης στο να θυμηθούμε ποιες ήταν οι αρχές της πολιτικής συνοχής, καλύτερα θα πρέπει ίσως να διαχειριστούμε την πολιτική συνοχή ώστε να λειτουργεί με καλύτερο τρόπο, να είναι πιο υποφελής Ακόμα θα πρέπει να είναι πιο, ε, προσβάσιμη η προσέγγιση των στα κονδύλια, η διάθεση των κονδυλίων, η προσπελασιμότητα σε αυτά οι όροι ε, λειτουργίας θα πρέπει να είναι κομμένοι και ραμμένοι ώστε να υπάρχει ε, αποδοτικότητα για τα κονδύλια που επενδύουμε. Θα πρέπει να επικαλύπτεται καλύτερα και να συντονίζεται καλύτερα με άλλες πολιτικές ή πολιτική συνοχή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, το γνωρίζω αυτό Πρόεδρε, αλλά για το θέμα των όρων και προϋποθέσεων ακούσαμε από αρκετού προλαλήσαντες παρατηρήσεις για τους όρους και προϋποθέσεις. Δεν είναι πραγματικά καθόλου καλή η συγκυρία χρονικά τους καιρούς που ζούμε και στην κρίση που περνάμε για να γίνεται λόγος για κυρώσεις και πρόστιμα τα οποία θα επιβάλλονται για τις χαμηλές επιδόσεις ή την κακοδιαχείριση από πλευράς κρατικών ή διοικητικών αρχών δίνει δυνατότητα αυτή η πολιτική προσέγγιση της πολιτικής συνοχής να υπάρχει μοχλικό αποτέλεσμα και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλα σχόλια και ερωτήματα, διότι επίτροπε το θέμα της μακροοικονομικής θέσης προποθέσεων πρέπει να το δούμε. Όμως να σας δώσω το λόγο σε πρώτη φάση, ε, γιατί σε εσά τέθηκαν τα περισσότερα ερωτήματα. Λοιπόν, είναι ευρύτερο το ζήτημα τη καλύτερη ε, επίτευξη αποτελεσμάτων. καλύτερου στόχου καλύτερο πολιτικό σχεδιασμό, ε, σαφή προστιθέμενη αξία. Ερωτήσεις, παρακαλώ, παρακαλώ. Ε, σηκώστε το χέρι σας, ναι. Ευχαριστώ. Ε, λέγομαι Ιβαν Ζάγκαρ και είμαι μέλος της Σλοβενικής Αντιπροσωπείας. Ε, πράγματι, η πολιτική συνοχή είχε σοβαρό ρόλο να διαδραματίσει στην ε, Σλοβενία εν των εξέλιξεων και για σκοπούς ανάπτυξης. Όμως, σε διαφορετικές χώρες υπάρχουν διαφορετικά συστήματα. Ως προς αυτό, λοιπόν, ήθελα να τονίσω ότι θα έπρεπε να αναζητήσουμε την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των μεγάλων προγραμμάτων μεν, αλλά και τα μικρότερα προγράμματα να μην τα παραγνωρίζουμε, διότι εκεί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σε συγκεκριμένου τομεί και εντό μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Και μία ερώτηση τώρα, περισσότερο είναι μια ιδέα που θα ήθελα να δώσω στο πάνελ. Είπατε τι ποσοστό του ΑΕΠ θα πρέπει οι χώρες να προβλέπουν για τις επενδύσεις στις περιφέρειες. Αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο ευρωπαϊκό, είναι και των εθνικών κυβερνήσεων. Είναι σαφές ότι το σύστημα παρά είναι άκαμπτο. Έχουμε βελτιωθεί, είμαστε πιο διαλλακτικοί, όμως η διαφορά μεταξύ μεμονωμένων περιφερειών πλέον σήμερα μπορεί να είναι τεράστια, μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσει πριν δώσω το λόγο στα μέλη του πανέλ. Επίτροπε, ακούσατε, ακούσατε ποια είναι η γενική αντίδραση. Ξεκίνησε η κυρία Μπρέσο λέγοντα ότι υπάρχει πολλή αυστηρότητα στην μακροοικονομική θέση προποθέσεων. Γιατί θα πρέπει να τιμωρούνται οι περιφέρειε λοιπόν για τα ασφάλματα των εθνικών κυβερνήσεων και αυτό πώ θα βοηθήσει τι χώρε που αγωνίζονται και γενικότερα μας ε, είπε και ο ε, συνάδελφος ότι γενικώ είναι πάρα πολύ οι όροι, πολύ ψηλά ο πύχης. Αλλά δεν είναι πολλά τα καρότα, είναι πολλά τα μπαστούνια. Λοιπόν, ίσως είναι περισσότερα τα μπαστούνια παρά τα καρότα. Απαντήστε μου εσείς και μετά η κυρία Μπρέσου. Um Για να μην υπάρξει μια τέτοια εντύπωση, δύο κράτη-μέλη αποστέλουν μια επιστολή και εμείς ε, να τρέχουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο τηλεφώνημα, η πρώτη κλίση που πήρα και δεν ήταν ακόμα επίσημο λόγω των μακροοικονομικών όρων και προϋποθέσεων ήταν από, μία από τις, ε, από ένα από τα κέντρα των κυβερνήσεων και δεν ήταν υποστηρικτικό τηλεφώνημα. Για να μην έχετε την εντύπωση ότι ένα προ ένα έχουν γίνει όλα δεκτά, καμιά φορά υπάρχει εντύπωση ότι υπάρχουν προτάσει ε, που θα ισχύουν για 26, 26 υπόλοιπου, αλλά όχι για τον εαυτό του. Στοχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υποβάλει προτάσει που θα ισχύουν και για τα 27 συνολικά κράτη-μέλη, χωρίς καμιά εξαίρεση. Για όλα μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά η απέτηση ήταν να μπορέσει να βρεθεί μια δυνατότητα, να υπάρχει μια δυνατότητα ως ultima ratio, δηλαδή ως έσχατη προσφυγή, δηλαδή να ισχύουν όλα ισότιμα για τα 27 κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις περιφέρειες τώρα, και αυτό σε σχέση με ένα κείμενο που αποτελεί συμβιβασμό και είναι αποτέλεσμα πολλών διαπραγματεύσεων και προσπαθειών και δεν είναι κάτι το ευανάγνωστο ακόμα και στη μητρική μας γλώσσα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτά τα οποία εμπεριέχονται λένε ότι αν και όταν φτάσει στην εφαρμογή αυτού του άρθρου η υπόθεση επιβολής προστήμων ή πίνων ε, έχουμε και ένα αντίστοιχο άρθρο του Ταμείου Συνοχής, στο Ταμείο δηλαδή Συνοχής, που ποτέ δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα και όχι επειδή δεν τολμήσαμε, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε αφορμή και αίτιο να γίνει αυτό. Αυτοί οι κανόνες τι λένε, αυτή η ρύθμιση τι λέει. Τα κράτη-μέλη, αν διαπιστωθεί ότι έχουν υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα και έχουν αποτύχει στο να πετύχουν τους στόχους ανάπτυξης, εδώ καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις και πρέπει να υποβάλει προτάσεις που θα λένε τι πρέπει να γίνει ώστε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση και να την θεραπεύσουμε, να την αντισταθμίσουμε. Αν τα κράτη-μέλη ανταποκριθούν σε αυτές τις προτάσεις μας και συμμορφωθούν, τότε δεν θα υπάρχει αφορμή και λόγος να καταλήξουμε σε αυτά τα μέτρα. Διότι πραγματικά το τονίζω, αυτά τα μέτρα είναι η αντιστάθμιση, η προσπάθεια επανόρθωσης και επιστροφής στη σωστή πορεία για τα κράτη που έχουν προβλήματα. Είναι σαφές ότι προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν συγκεκριμένα μέσα. Μόνο όταν υποτροπιάζουν κράτη-μέλη και επανειλημμένα αρνούνται να συμμορφωθούν και να ευθυγραμμιστούν, ε, τότε για τα λειτουργικά προγράμματα τα οποία σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής τους και προσαρμογής τους που πρέπει να υιοθετηθεί δεν γίνεται τίποτα από τα κράτη-μέλη αυτά πρέπει να υπάρχει ως έσχατη προσφυγή ένας μηχανισμός κυρώσεων και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους εκπροσώπους των περιφερειών υπάρχει αυτή η ρύθμιση ότι αναλογικά θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο αν και όταν χρειαστεί να εφαρμοστεί σε περιφέρειες που έχουν υψηλή αυτονομία και δεδομένη αυτονομία και είναι αυτοτελείς ή αυτούσιες δεν να φανταστώ, να φανταστώ ότι λειτουργικά προγράμματα για αυτές τις περιφέρειες θα πληγούν. Δεν συμβαίνει ότι αυτόματα όλα τα προγράμματα σε πλήρες ε, μέτρο και εύρος θα είναι αντικείμενα κυρώσεων και προστήμων κάποια προγράμματα θα μπορεί να είναι αυτά. Και μέσα στο πλαίσιο αυτών των κάποιων συγκεκριμένων προγραμμάτων θα πρέπει να υπάρχει ύψος αναλογικής εφαρμογής της ποινή ή της κύρωσης όσον αφορά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την λέξη ποινή, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω την λέξη εφαρμογή μ, συμμόρφωσης. Ευχαριστώ. Και για το επιχείρημα ότι είναι πολλά τα μπαστούνια και λίγα τα καρότα, τι λέτε. Uh, Γι' αυτό συζητούμε μόνο τα μπαστούνια και τα καρότα για την ώρα. Τέλος πάντων, ο κύριος Σνάιντερ νομίζω είπε, καθώς και κάποιοι άλλοι, ότι το 90-95% των προτάσεων εγκρίνονται, βρίσκουν σύμφωνους τους ε, υπευθύνου. Τώρα το 5% μπορούμε να το συζητήσουμε. Μας απασχολεί συνήθως ένα πεντάλεπτο το πολύ, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτή ήταν η γενικότερη εικόνα και θέμα τη συνολική πρόταση. Μάλιστα, ε, όμω ο Μισελ Τελαμπάρ μα είπε για δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι των ε, περιφερειών. Όχι, είπατε ότι είναι λύση η τελευταία επιλογή ε, να ανατρέξουμε στα κράτη-μέλη. Τελικά το αποδέχεστε έστω και λίγο το επιχείρημα ότι η αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής ε, επηρεάζεται από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Υπάρχει διασύνδεση, δεν χρησιμοποιείται ως ε, εργαλείο ή όπλο για να τιμωρηθούν ε, κάποιοι για το σφάλματο στον άλλο τομέα. Ναι, μου λέτε αν το οικονομικό περιβάλλον είναι κακό, μήπως κλείνουμε την κάνουλα και μήπως πρέπει να κλείσουμε και το κατάστημα της πολιτικής συνεχής και να πάμε σπίτια μας. Βεβαίως χρειάζεται και με καλό μικροοικονομικό περιβάλλον για να ευδοκιμήσει η πολιτική συνοχής. Γι' αυτό κάποιες φορές και παίρνουμε κονδύλια. Εάν ε, δεν λειτουργεί μακροοικονομική βέβαια πολιτική δεν θα σωθεί από την πολιτική συνοχής και τα κονδύλια της. Όμως ε, πριν από ένα χρόνο, όταν πρώτη φορά ακούστηκε αυτή η ιδέα, εγώ αντιτάχθηκα και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε τα μακροοικονομικά με το Ταμείο Συνοχής, διότι σκοπός του είναι να διευκολύνει την ε, ε, διευκόλυνση της νομισματικής ένωσης. Αυτό προβλέπεται από τη συνθήκη τέτοια διασύνδεση με τις μακροοικονομικές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικό πράγμα, γι' αυτό και εγώ φρόντισα να διαχωρίσω τη θέση μου. Τώρα, το αν είναι λογικό να τιμωρούμε μέσω, μέσω των εργαλείων που μας διατίθενται μέσω άλλης πολιτικής για το τι συμβαίνει σε έναν άλλο πολιτικό τομέα. Βεβαίως, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό εκτός του κάθε πολιτικού τομέα, στα πλαίσια τη ίδια τη πολιτική πρέπει να αναζητούμε τα σφάλματα. Αλλά σκεφτούμε την Ελλάδα που έχει αυτή τη στιγμή τόσα προβλήματα. Και κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα και με τα διευθυντικά ταμεία και με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συνοχή γενικότερα. Λοιπόν, δεν μπορεί να βρούμε τώρα ένα άλλο μέσο που να αντιτίθεται σε αυτή τη λογική. Επίση, ε, ελπίζω ότι με τα επιχειρήματα που τέθηκαν και ήταν τόσο πολλαπλά να έχετε μια ζωή συζήτηση για όλα αυτά. Είναι δύσκολο να βγάλουμε ένα οριστικό συμπέρασμα σήμερα, όμω πρέπει να σκεφτούμε όλε τι προοπτικέ και να δούμε κατά πόσον υπάρχουν τιμωρίε και μπαστούνια, όπω λέτε, στην πολιτική συνοχή ή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εμεί θέλουμε στην πολιτική συνοχή, με μια σειρά από τιμωρίε, να καταφέρουμε τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τα διαθέσουμε στι περιφέρειε τελικά. Δηλαδή, ούτω ή άλλω. Δεν θα πρέπει να ακούμε τα αντίθετα επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν. Ε, σα ευχαριστώ και θα ήθελα την αντίδρασή σα για αυτά που ακούσατε για τι μακροοικονομικέ περιστάσει. Τι είναι το καλύτερο, τα μπαστούνια, τα καρότα θα δεχτείτε το επιχειρήμα της Επιτρόπου, του Επιτρόπου ότι το 5%, είναι, το 5 είναι το θέμα είναι το κριτήριο των επιδόσεων. Είναι μεγάλο το καρότο. Μήπω πρέπει να το σκεφτούμε τελικά από την άποψη των όρων και όχι των ανταμοιβών. Πιστεύω ότι λειτουργεί καλά το μπαστούνι και το καρότο. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Δεν είναι το όργανο αυτό το οποίο μπαίνει στο καθεστώς ε, του μπαστούνιου. Η πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική επενδύσεων μακροπρόθεσμα, η οποία επιτρέπει πρώτα απ' όλα στις χώρες και μετά στις περιφέρειες που είναι οι δικαιούχοι στις περισσότερες χώρες των κονδυλίων αυτών, να προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα την πολιτική τους επενδύσεων. Σήμερα 65% των δημοσίων επενδύσεων στην Ευρώπη γίνεται από τις περιφέρειες και την τοπική αυτοδίκηση. 65% έτσι. Ενώ μόνο το 15% του χρέους αφορά την τοπική αυτοδίκηση. Οπότε αν σκεφτούμε ότι με αυτή τη δαμόκλειο σπάθη θα μπορούσαμε να δουλέψουμε καλύτερα, ε όχι, διαπιστώνουμε πως δεν είναι αλήθεια. Διότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις επενδύσεις μαζί μας θα έχουν την ανησυχία ότι ξεκινάνε μια μακρά διαδικασία επενδύσεων χωρίς να είναι σίγουροι ότι θα αποδώσουν τα χρήματά τους στο τέλος. Και προσθέτω και κάτι ακόμα. Η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στην Επιτροπή των Περιφερειών το καθήκον της στήριξη της επικουρικότητας και μάλιστα μας έδωσε το δικαίωμα να φτάσουμε και με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το μελετήσαμε το θέμα γιατί είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση όπου δεν επιλέγουμε το σωστό θεσμικό όργανο που το βάζουμε κάτω από το μικροσκόπιο. Οπότε είναι απόλυτα λογικό να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας και αναλογικότητας. Διότι βέβαια και είναι σωστό ότι πρέπει μια περιφέρεια η οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει καλά ε, τους πόρους της πρέπει να τιμωρηθεί. Αυτό το δεχόμαστε και το θέλουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να τιμωρούμε κάποιον ο οποίος πολύ πιθανό να μην έχει καμία ευθύνη. Αν λοιπόν μου πείτε, στην περίπτωση που και οι περιφέρειες είναι χρεωμένες, δεν τηρούν το συμφωνό σταθερότητα, το παραβιάζουν, για τα δικά τους δημοσιονομικά σύμφωνοι. Αλλά προσοχή, είδαμε στις περιφέρειές μας ότι όταν μακροχρόνιες επενδύσεις ξαφνικά σταματάνε, τότε είναι που δεν μπορούμε πια να μιλάμε για ανάπτυξη. Και αυτή είναι η ανησυχία μας. Το γεγονός δηλαδή ότι κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική επιπλέον στους επενδυτές οι οποίοι ήδη είναι ανήσυχοι και ήδη δυσκολεύονται να επενδύσουν. Πόσο μάλλον. Κυρίε και κύριοι, δεν θα το λύσουμε το θέμα τώρα. Οι διαπραγματεύσει και σκληρέ θα είναι και μακρέ. Τέλο πάντων, η Επιτροπή είναι έτοιμη για μάχη. Α περάσουμε τώρα στο τρίτο μα ζήτημα για σήμερα το απόγευμα, η γεωγραφική διάσταση. Η Υπουργό Μπιενκόφσκα το υπογράμμισε ιδιαίτερα στην παρουσίαση τη. Γιατί η εδαφικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι τόσο σημαντικά στον εντοπισμό των περιφερειών και των αναγκών τους ε, και μέσω των νέων προτάσεων. Α το δούμε λοιπόν, ας δούμε και το επόμενο φιλμάκι μας πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Dr. Sabo, please. Ε, είναι τελωνιακό, λέγομαι Λάζιλο και το γραφείο μου βρίσκεται στο Μόχατ στην Ουγγαρία. Είμαι υπεύθυνο για τον έλεγχο πολιτών και αγαθών που περνούν από το Δούναβι. Για μένα το σύστημα Νεβάντα ε, βελτιώνει τις επιδόσεις μου και μου παρέχει πιο σύγχρονες συνθήκες και δυνατότητες. Χάρη την καταγραφή των θέσεων των σκαφών μπορούμε να προετοιμαστούμε από την τελωνιακή την πλευρά για να δούμε ποιοι πάνε να διασχίσουν τα σύνορα και να έχουμε καλύτερη φύλαξη των σύνορων. Με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν η ροή των πληροφοριών μέσω των σερβικών, κροατικών και ουγγρικών σύνορων είναι πιο αποτελεσματική. Okay. Πολύ ωραία. Τώρα βλέπουμε πώς ένα από τα στοιχεία του νέου νομοθετικού πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει τις ε, περιοχές όπως αυτή τη Δούναδη που είδαμε αλλά και στη Βαλτική θάλασσα. Να δούμε λοιπόν ποιοι ζήτησαν το λόγο από την αρχή. Ο κύριος Καμίνης, σύνορχος της Αθήνας, μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών. Παρακαλώ. Ακούγομαι. Κυρίες και κύριοι, παρόλο που όλοι σχεδόν οι προηγούμενοι ομιλητές δεν προέρχονται από χώρες που έχουν πληγεί βαριά από την κρίση, όλοι τους εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στις τοπικές και περιφερειακές αρχές των χωρών αυτών που είναι αντιμέτωπες, θα έλεγα, με μια ουσιαστικά σχεδόν υπαρξιακή κρίση και πολλοί είναι αυτοί που εκφράστηκαν εναντίον της μακροοικονομικής συμμόρφωσης στη μελλοντική περιφερειακή πολιτική. Θα ενώσω και εγώ τη φωνή μου με αυτούς, αλλά θα μιλήσω και για τα καρότα. Δεν θα μιλήσω μόνο για τα βαστούνια. Θα ήθελα περισσότερο να εστιάσω στις αστικές περιοχές, εντάσσοντας βέβαια στο ευρύτερο πλαίσιο της γεωγραφίας και όταν λέμε γεωγραφία πια θα πρέπει όταν αναφερόμαστε στην πολιτική συνοχής να μην σκεφτόμαστε μόνο με όρους της κλασικές αυτές διαφοροποιήσεις που γνωρίζουμε μεταξύ Βορρά-Νότου, Ανατολής-Δύσης ή και ακόμη μεταξύ των χωρών που είναι καθαρά εισφορείς και των χωρών που είναι καθαρά αποδέκτες. Η γεωγραφία συνιστά ουσιαστικά μια δεύτερη διάσταση της πολιτικής ε, της συνοχής μια δεύτερη διάσταση που λαμβάνει υπόψη ολοκληρωμένες εδαφικές προσεγγίσεις με βάση τη γεωγραφική ιδιωτερότητα και προωθούν λύσεις που εμπλέκουν διαφορετικούς τομείς, διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης και που είναι συχνά εξαιρετικά καινοτόμες. Ειδικά οι προτάσεις για τις αστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορώ να πω ότι υπερβαίνουν σοβαρές προσδοκίες Ελπίζω ειλικρινά να μείνει σταθερά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμείνει στις προτάσεις της που αφορούν τις αστικές περιοχές και να αντισταθεί σε όλους αυτούς που θα θελήσουν να αμφισβητήσουν τα φιλόδοξα σχέδιά της υπό το πρόσχημα ότι δεν υπάρχει σαφής νομοθετική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πολιτικής για τις αστικές περιοχές. Οι πόλεις επηρεάζονται άμεσα από πάρα πολλές πολιτικές της Ένωσης όπως αυτές που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες, <clears throat> τις μεταφορές, το περιβάλλον και την ενέργεια. Οι πόλεις είναι ατμομηχανές της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και μια ιδιαίτερη πρόκληση για τη συνοχή. Αυτό γιατί πίσω από τις εντυπωσιακέ στατιστικές που αφορούν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των αστικών περιοχών, πάρα πολύ συχνά, κατά κανόνα μάλλον θα έλεγα, υπάρχει μια άλλη λιγότερο λαμπερή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που αποτυπώνεται με άλλους δείκτες και όχι μόνο μέσω του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η κρίση πλήττει πρώτα απ' όλα τις αστικές περιοχές, στις προηγμένες τουλάχιστον οικονομικά χώρους και κατά δεύτερο λόγο τις αγροτικές. Επικροτούμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσει την πολιτική για τις αστικές περιοχές οριζόντια στην πρότασή της για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και σε αυτήν για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η λέξη αστικός επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στις 11 προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τις μεταφορές, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της φτώχειας. Και είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι επιβάλλεται ένα 5% της χρηματοδότησης για αστικές περιοχές σε κάθε κράτος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κάποιες ερωτήσεις για τον Επίτροπο πώς θα αλληλοεπιδράσει η επωνομαζόμενη πλατφόρμα ανάπτυξης αστικών περιοχών τελειώνω με τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συμφώνου των Δημάρχων ή με τις πρωτοβουλίες για τις έξυπνες πόλεις. Ποια θα είναι η συσχέτιση μεταξύ της πλατφόρμας ανάπτυξης αστικών περιοχών και της δέσμης γάμα του νέου προγράμματος Ίντερεγ. Και τέλος, the και τέλος γιατί επιλέξατε να ορίσετε το ανώτατο όριο αντί για το κατόφλι για καινοτόμε δράσει στο ύψο του 0,2 τη συνολική ετήσια εκχώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ρομινάρο. Τώρα, περιφερειακό Περιφερειακός Υπουργός για την Εκπαίδευση και την Καινοτομία στην Γουλή Βενέτσια και Τζούλια, Ιταλία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώ το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας μιας αυτόνομης περιφέρειας βορειοανατολικά της Ιταλίας. Είναι διασυνοριακή περιοχή και στο κέντρο της σημερινής Ευρώπης. Η διασυνοριακή συνεργασία για μας βρίσκεται στο DNA μας. Αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της διασυνοριακής μας κοινότητας, η οποία επέτρεψε να κρατήσουμε ανοιχτό το διάλογο με τις χώρες του τέο μπλοκ, ακόμα και κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα πώς θα βγούμε από την κρίση. Και θα βγούμε από την κρίση μόνο με συνεργασία. Υπάρχουν όμως και άλλες ανησυχίες σήμερα εν ώψη του 2020 και αυτές έχουν να κάνουν με το μέλος της πολιτικής συνοχής. Στις περιφέρειές μας η πολιτική συνοχής έχει μια προστιθέμενη αξία γιατί βοηθάει στην ανταγωνιστικότητα. Οι αυτοματισμοί δεν είναι ικανοποιητικοί. Θέλουμε ελαστικότητα στην εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής. Μόνο με μια βιώσιμη δράση στην οποία συμμετέχουν όλοι υπέρ της εκπαίδευσης και της μόρφωσης μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Να για μας ποια είναι η προτεραιότητα. Και από εκεί και πέρα εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόταση της Επιτροπής που θέλει να διατηρήσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας, ε, να το προχωρήσει μετά το 2013 πολύ περισσότερο, όπως επίσης και η ιδέα για μια κεντρική υπηρεσία που θα ασχολείται με τις διασυνοριακές περιοχές. Εμείς θέλουμε σύνδεση με τα πανεπιστήμια, γιατί είναι κάτι που μπορεί να έχει Επιπτώσει στην επικράτεια. Με συγκεκριμένε δράσεις λοιπόν και συνεργασία με τα πανεπιστήμια στις διασυνοριακέ περιοχές πιστεύω ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε. Σκέφτομαι τώρα το δίκτυο του Δούναβη, της Αδριατική. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα, υπάρχει δυναμικό προκειμένου να αναπτύξουμε μια κοινή γραμματεία στα πλαίσια της αντιπροσωπείας μας στις Βρυξέλλες. Και στρέφομαι προς τον Επίτροπο για να στηρίξει ακόμα περισσότερο την πρόταση της Επιτροπής και στην κυρία Χίμπνερ για να της πω ότι θα παίξουμε το ρόλο που μας πρέπει σε περιφερειακό επίπεδο για να έχουμε μια πολιτική συνοχής η οποία θα μας επιτρέψει με τις ε, γείτονες χώρες τις πιο πρόσφατες αλλά και τις μελλοντικές, να έχουμε μια πολιτική συνοχής που να είναι αντάξια των στόχων του 2020. Ο Χέσους Καμάνο Αλεπίσης έχει τώρα το λόγο από την Γαλλικία, Ισπανία, μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών και συγητής για τον κανονισμό για το Ιωρικό Ταμείο. Πού είσαστε? Να σας δούμε. Εκεί, ναι. Είναι πολύ μεγάλη αίθουσα. Τώρα σας είδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντέβης. Είναι προφανές, όπως είπε και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ότι η οικονομική και η δημοσιονομική κρίση δεν επηρεάζει εξίσου όλες τις περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική και η δημοσιονομική κρίση όμως στην Ευρώπη ε, πρωταγωνιστεί στη συζήτηση σήμερα για παράδειγμα το απόγευμα. Δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικό γιατί απαιτήθηκαν μέτρα λιτότητας και οι περισσότερες χώρες επέβαλαν μέτρα στα οποία πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι οι πολίτες. Πρέπει εδώ να πω ότι αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τέτοιες δυσκολίες, το περιφερειακό επίπεδο, οι περιφέρειες παίρνουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί ακριβώς εκεί είναι που φαίνεται ότι η εδαφική συνοχή είναι πραγματικά μια δημοκρατική συνοχή, μια πολιτική δηλαδή που επηρεάζει όλες τις περιφέρειες και που μπορεί να ερμηνευτεί όχι μόνο σε σχέση με τις δαπάνες αλλά και σε σχέση με τις επενδύσεις. Άρα λοιπόν απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών προκειμένου να χρησιμοποιούμε τους λίγους πόρους που έχουμε. Η στρατηγική για το 2020 συνεπώς σημαίνει ότι η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε την αηφόρο ανάπτυξη με στρατηγικές που υπακούν σε κοινέ αρχές. Συνεπώς, ό,τι ευρωπαϊκή συνεργασία υπάρχει, η ICT, για παράδειγμα που αποτελούν σημαντικό μέσο για το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας, της διαπεριφερειακής στην Ευρώπη, είναι κάτι που έχει να παίξει σημαντικό ρόλο διότι φτιάχνουν δίκτυα συνεργασίας και διαλόγου γιατί επιτρέπουν να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές και γιατί προχωρούν ε, προγράμματα ανάπτυξης. Επίσης αποτελούν βασικό στοιχείο καθορισμού της περιφερειακής πολιτικής επιτρέποντας δομές συνεργασίας σε διασυνοριακό επίπεδο και καθορίζουν και στρατηγικές ανάπτυξης, όπως επίσης δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, διαχειρίζονται προγράμματα και κοινού πόρους. Ολοκληρώνω κυρία Ντέιβις με το εξή. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι έλαβε υπόψη της κάποιες από τις συστάσεις του ψηφίσματος που ενέκρινε η Επιτροπή των Περιφερειών για τις Ευρωπαϊκές ε, Ομάδες Συνεργασίας. Ακούσαμε τον κύριο Μπαρόσο σήμερα που είπε ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα μέσα της πολιτικής συνοχής. Πιστεύω και το λέω αυτό στον Επίτροπο Χαν ότι χρειάζεται και περισσότερη ε, στήριξη στη διασυνοριακή συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο της εδαφικής συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει περάσει κάπως ο χρόνος, αλλά υπάρχει κάποιος πηγόντος που έχει να πει κάτι πριν να επιστρέψω στο πάνελ. Γιατί θέλω και το πάνελ να μπορέσει να πάρει το λόγο. Κάτι καυτό. Εσείς, πολύ σύντομα, παρακαλώ. Καστιλιώνη από την Κατάνια. Από την Κατάνια, πρόεδρος ε, των ε, περιφερειών των επαρχιών στην Ιταλία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και την, τον, την Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έδωσαν πολύ μεγάλη προσοχή στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και ο Επίτροπος Χάν έτεινε βίκονούσα, άκουσε προσεκτικά φουγκράστηκε τις προτάσεις μας και δεν γίνεται μόνο αναφορά σε σχέση με αυτά τα βιντεάκια, πρόκειται για σύντομες αναφορές. Υπάρχουν όμως περιφέρειες που έχουν αρκετά κονδύλια όσον αφορά τα, την α, χρήση τους, όμως υπάρχουν προβλήματα απορροφητικότητας και προβλήματα απορρόφησης κονδυλίων. Υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία έχουν περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα, είναι περισσότερο πολιτικά ζητήματα. Θα ήθελα να πω στον Επίτροπο Χάν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την άμεση συμμετοχή, σε σχέση με την χρήση των κονδυλίων των διαθετικών ταμείων, υπαναχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια θα είναι στο μέλλον. Θα είναι περισσότερη η εμπλοκή της Επιτροπής ή θα είναι συμπληρωματικός και παραπληρωματικός ο ρόλος της. Γνωρίζουμε ότι από πλευράς ε, της συνεργασίας μεταξύ εθνικών προϋπολογισμών και ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα έπρεπε να υπάρχει ένας, ε, μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση στο συντονιστικό αυτό ρόλο ή θα, υπαναχωρεί, θα υποχωρεί η θα ειναι συμπληρωματικος και παραπληρωματικος ο ρολος της γνωριζουμε οτι απο πλευρα της συνεργασιας μεταξυ εθνικων προυπολογισμων και ευρωπαικου προυπολογισμου Επιτροπή και στο τέλος τέλος ε, θα βρίσκεται πίσω από συγκεκριμένες γραμμές τεράστια θέματα αυτά όσον αφορά τα αστικά κέντρα της πόλης μας. Ε, πρέπει να δούμε τις υποδομές και πρέπει να επενδύσουμε στην κινητικότητα, στην ενέργεια, στο ευρύ, ε, φάσμα ε, συχνοτήτων όσον αφορά τα πιο φλέγοντα θέματα παρέμβασης ε, αν είναι δυνατόν θέλετε να πείτε κάτι όχι εντάξει λοιπόν για οποιαδήποτε δυνατότητα τοποθέτησης πρωτού κλείσουμε αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να προσπαθήσουμε να ταυτοποιήσουμε κάποιες προτεραιότητες να συζητήσουμε ευρύτερα για το θέμα των ανοιχτών ημερών επενδύοντας το μέλλον της Ευρώπης πόλεις και δίνοντας πρόσθετη αξία. Είναι ένα πακέτο μέτρων. Πώς θα συνεισφέρουμε, πώς οι εκπρόσωποι σε, αυτό, σε αυτή την αίθουσα, οι πόλεις, οι περιφέρειες θα μπορέσουν να συνεισφέρουν σε σχέση με τις τελικές ε, παρατηρήσεις σας. Αν έπρεπε να ε, ταυτοποιήσετε μια κύρια προτεραιότητα που θα μπορούσε να βοηθήσει να επιτύχουν οι πόλεις και οι περιφέρειες, ποια θα ήταν η ανώτατη προτεραιότητα από τα πολλά θέματα τα οποία αναβέθηκαν και καλύφθηκαν. Με άλλα λόγια δηλαδή, είπατε στην αρχή κυρία Χούμπνερ, η πολιτική συνοχή είναι πολιτική δημιουργία εμπιστοσύνη. Τι θα έδινε την μέγιστη εμπιστοσύνη ω μέτρο ή ω πρωτοβουλία, τι θα βοηθούσε τι πόλει και περιφέρειε περισσότερο. Εσεί ε, πρώτα, κυρία Μπρέσο, μετά η Επιτροπή και μετά η κυρία Χούμπνερ για να ολοκληρώσει. Λοιπόν, παρακαλώ να απαντήσετε και στα σχόλια που έγιναν ε, προηγούμενα σε σχέση με την καταληκτική αυτή τοποθέτησή σας. Η κυρία Μπρέσο, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ η ίδια αν έπρεπε να προσδιορίσω ένα στοιχείο, ένα παράγοντα, είναι πολύ δύσκολο βέβαια να επιλέξει κανείς ένα και μόνο. Θα έλεγα η πολιτική για τα ενεργειακά θέματα, η ενεργειακή πολιτική θα βρισκόταν μάλλον στο επίκεντρο της ε, πολιτικής για την καινοτομία από πλευρά μας τα επόμενα χρόνια, στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής. Αυτό αληθεύει για πολλές ε, περιφέρειες και σε σχέση με την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και τη δέσμευσή μας ε, να κάνουμε κάτι, να διασφαλίσουμε την αηφορία στις περιφέρειες και στο πλαίσιο των τοπικών αρχών. Νομίζω συμφωνούμε όλοι για την σημασία που έχουν τα ενεργειακά ζητήματα και αυτό μου επιτρέπει να επιλέξω να αναφερθώ σε ένα αίτημα που εκφράστηκε από πολλούς. Αληθεύει ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την πολιτική μας για τα αστικά κέντρα και τις πόλεις. Ολοκλήρωση, κινητικότητα ευφυής, ε, ανάπτυξη, αηφόρος ανάπτυξη Κάνοντας λόγο για όλα αυτά πρέπει να δούμε τι γίνεται στα αστικά κέντρα και στις πόλεις μας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν στις πόλεις μας και στα μητροπολιτικά κέντρα και πρέπει με τις σωστές ιδέες να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε. Και όσον αφορά και το τελευταίο θέμα το οποίο αφορά την κοινωνική συνοχή και τα μέσα και εργαλεία για να προωθεί η κοινωνική συνοχή θα έλεγα ότι σήμερα ουσιαστικά πράγματι είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Χάν για τους νέους κανονισμούς και διατάξεις και είδαμε και τα διάφορα προγράμματα τα οποία λειτουργήσαν τα τελευταία χρόνια. Το θέμα της ε, περιφερειακής συνοχής ως ζήτημα είναι ένα θέμα που δίνουν τεράστια σημασία σε αυτό οι περιφέρειες η συνοχή έχει τεράστια σπουδαιότητα. Μπορούν να συνδυαστούν ε, οι νέοι στόχοι με την απλούστευση και την χρήση των ε, ε, μέσων αυτών. Μία από τις ιδέες είναι να χρησιμοποιηθούν δίκτυα, η δικτύωση ως μέσα, ως εργαλεία για να δημιουργηθεί μία μάκρο περιφερειακή προσέγγιση όχι μόνο για την περιοχή του Δούναβη, της λεκάνης του Δούναβη, ούτε μόνο για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Υπάρχουν και άλλες ευρύτερες μακροπεριφερειακές δυνατότητες προσέγγισης περιφερειών σε μια ενοποιημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε με τη χρήση αυτών των νέων μέσων. Είναι φυσικά πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί ε, η σωστή περιφερειακή συνοχή ε, στην Ευρώπη συλλήβδην. Πρέπει να ταυτοποιήσουμε περιφέρειες ως ε, ε, θα έλεγα ενώσεις μέσα σε ένα μεγαλόπνο σχέδιο, μέσα σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κύριε Χαν, αν έπρεπε να δείξετε ένα θέμα, δεν ξέρω αν θα πείτε εσείς ότι είναι οι προϋποθέσεις, θα ήσασταν πολύ θαραλέως να το κάνατε. μάκρο και μικρο είναι πάντα μια διαφοροποίηση. Θέλω πρώτα να ζητήσω συγγνώμη για εκείνους που δεν μπόρεσα να αναφερθώ και να υπησέλθω στις παρατηρήσεις και ερωτήσεις τους. Όμως από πλευράς Ντέιβις υπήρξε ένα αυστηρό καθεστώς διαχείρισης ε, των συζητήσεων. Θα πρέπει να δραχθούμε των ευκαιριών τις επόμενες ε, ημέρες. Υπάρχουν πολλοί συνεργάτες που βρίσκονται καθοδόν για να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα ή θα προσπαθήσουμε γραπτός να σας απαντήσουμε αν όχι διμερός, για την ιδιαίτερη πρόθεση των ορεινών περιοχών. Κάθε περιφέρεια μέσα στο πλαίσιο της θα πρέπει να έχει δυνατότητες ποσοστώσεων συγχρηματοδότησης και διαμόρφωσης αυτών των δυνατοτήτων και να θέσει ίδια η περιφέρεια κέντρα βάρους. Δεν παρακολείται, δεν υπάρχει παρεμπόδιση κάποιας περιφέρειας να χρησιμοποιήσει κονδύλια σε μεγαλύτερο ποσοστό ή και σε συγχρηματοδότηση ή και για ένα άλλο τμήμα, για ένα άλλο μέρος αυτής της περιφέρειας διαφορετικά, διαφορετικά ποσοστά χρηματοδότηση. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για τις εξατομικευμένες δυνατότητες προσέγγισης και δράσης που έχουμε αναφέρει. Αν με ρωτάτε ποια είναι η ανώτατη προτεραιότητα, θα έλεγα η πολιτική είναι για να είναι διάκριτα τα αποτελέσματα της δράσης μας για τους πολίτες μας να δουν ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν είναι ε, κάποια, ε, κάποιος κενός λόγος, αλλά ότι η Ευρώπη είναι σε θέση με τους πολίτες της να δημιουργήσει πρόσθετη αξία και με αυτές τις δράσεις ε, να δώσει θετικά αποτελέσματα. Να δούμε με μια συνεκτική προσέγγιση για την ενεργειακή πολιτική, για παράδειγμα, ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να επιτευχθεί και να μπορέσουμε να έχουμε μια προσέγγιση και για την μακροπεριφερειακή επικέντρωση, τον μακροπεριφερειακό εστιασμό. Να είμαστε μέσα σε ένα διαφανές πλαίσιο αποτελεσματική για τους πολίτες της Ευρώπης. Να βλέπουν ευδιάκριτα ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα των δράσεών. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χούμπνερ προκειμένου να πάρει το λόγο και να καταλήξει αλλά προηγουμένως να απαντήσει σε ερωτήσεις. Θέλετε να τα κάνετε μαζί ή χωριστά. Καλά, πρώτα απαντήστε, μετά δώστε μου το λόγο και μετά πάλι θα σας το δώσω. Νομίζω Κοιτάξτε, λέμε καμιά φορά τα λεφτά δεν ε, πειράζουν. Όχι. Αυτή τη φορά δεν μπορούμε να λέμε κάτι Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα λεφτά δεν έχουν σημασία. Όχι. Και το είπαν και όλοι οι συμμετέχοντε ότι για να είναι αποτελεσματικέ επενδύσει, αυτό ακριβώ είναι που λέει και ο Επίτροπο Χάνο ότι θέλει. Δηλαδή να υπάρξει αρκετή χρηματοδότηση. Και όχι μόνο σε επίπεδο κοινοτικού προπολογισμού, αλλά και στι μικρέ περιφέρειε, στι πόλει, κινδυνεύουν να μην έχουν αρκετά χρήματα για να ξεκινήσουν προγράμματα να λύσουν τα προβλήματά τους. Αυτό λοιπόν που εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από όλους εμάς. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να καταλήξουμε στο καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν εξαρτάται όμως από εμά. Έχει να κάνει με το τι χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό, το πόσα χρήματα έχουμε. Ακόμα κι αν η πολιτική συνοχή δεν είναι μόνο χρήματα, τη συνοδεύουν ένα σωρό αξίες, θεμελιώδεις. Και αν θέλετε να περάσω στις παρατηρήσεις που είχα να κάνω για να κλείσουμε τη σημερινή μέρα. Να συνοψίσω είναι δύσκολο. Είπατε τόσα πολλά και σοφά πράγματα με τόσο ωραίο τρόπο, δύσκολα θα συνοψίσω. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δείξατε ε, και επιδείξατε υψηλό αίσθημα ευθύνης και θέλω επίση να σα επιβεβαιώσω για τη δικιά μα δέσμευση να δουλέψουμε υπέρ τη επιτυχία των στόχων τη στρατηγική 2020. Και ο Επίτροπο Χάν και εγώ και η κύριε Μπρέσο δεν νιώθουμε μόνοι μα. Ξέρουμε ότι έχουμε όλου εσά στο πλευρό μα. Αυτό το οποίο φάνηκε από τα σχόλιά σα είναι ότι επιβεβαιώνεται ότι συμφωνείτε μαζί μα πως η ανάπτυξη πρέπει να έρθει από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, από τις επιχειρήσεις, από όλους αυτούς που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και απασχόληση. Ο δικός μας ο ρόλος εδώ των θεσμικών οργάνων είναι να βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας στην υπηρεσία της επιτυχίας των στόχων. Και νομίζω ότι μιλάω εκ μέρους όλων εδώ. Αυτό θα το κάνουμε. Πιστεύω επίσης ότι αυτό που προσπαθήσατε να μας πείτε είναι ότι η πολιτική αυτή πρέπει να συνεχίσει να κάνει περισσότερα εκεί που υπάρχει κάποια καθυστέρηση, εκεί που υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Όμως η πολιτική αυτή πρέπει να υπογραμμίσει και τις περιοχές εκείνες όπου εντοπίζονται νέες δυνατότητες, νέες ευκαιρίες. Να ληφθεί υπόψη δηλαδή η διαφορετική κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των περιφερειών και των πόλων περιφερειακή συνοχή, είπαμε, και ο ρόλος των τοπικών αρχών. Αυτό είναι επίση κάτι που ακούστηκε πολλές φορές σήμερα στη συζήτηση. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου για το ότι η εδαφική συνοχή δεν αποτελεί έναν αυτοσκοπό, δηλαδή δεν είναι επειδή το λέει η συνθήκη ότι πρέπει να πετύχουμε την εδαφική συνοχή. Από αυτά που είπατε, εγώ κατάλαβα ότι αυτή η εδαφική συνοχή αποτελεί ένα μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και καλύτερη ανάπτυξη. Σημαίνει συγχρόνως ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να πετύχουμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που θα έρθουν από πάνω προς τα κάτω και σε αυτά που θα έρθουν από κάτω προς τα πάνω. Θέλω επίσης, έχοντας ακούσει όσα είπατε για τις κυρώσεις, για τα μπαστούνια και τα καρότα, ότι όλοι συμφωνούμε πως δεν θέλουμε το μέλλον της Ευρώπης να βασιστεί σε αυστηρές ποινές. Η μακροοικονομική αιρεσιμότητα πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν άδικη και παραγωγική. Αν σταματήσει η χρηματοδότηση αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στις περιφέρειες. Ενώ στην πραγματικότητα ε, είναι για να τιμωρηθεί η κακοδιαχείριση σε κεντρικό επίπεδο. Αυτά τα μέτρα λοιπόν αιρεσιμότητας θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την πολιτική συνοχής και ε, να υπάρχει πάντα διάλογος ανάμεσα στην ε, Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Δεν το συζητήσαμε τώρα πολύ, αλλά νομίζω ότι η απλοποίηση είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και δεν πρόκειται μόνο για τις διαχειριστικές αρχές, για το σύστημα που διαχειρίζεται την πολιτική αυτή, έχει να κάνει και με τους ίδιους τους δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν λιγότερη γραφειοκρατία να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα, επειδή η πολιτική μας προσανατολίζεται στα αποτελέσματα, είναι κάτι που όλοι θέλουμε. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε περισσότερες προσπάθειες στην ε, ε, μεταφορά των αποτελεσμάτων, αλλά η ενέργειά μας να δοθεί στα ίδια τα αποτελέσματα, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όταν είπαμε ότι ευθυγραμμίζουμε την πολιτική μας με τους στόχους της στρατηγικής του 2020 και επικεντρώνουμε τους πόρους μας σε ένα περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, να ξέρετε ότι μας απασχολεί πάρα πολύ η ευαισθησία που δείχνουν οι περιφέρειες. Γι' αυτό η αρχή αυτή δεν θα πρέπει να πλήξει τις περιφέρειες που έχουν ανάγκη αποστήριξη. Και θέλω επίσης να σας πω ότι για άλλη μια φορά για τη χρηματοδότηση πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το εξή. Και αυτό το κατάλαβα από αυτά που είπατε και είναι και η δικιά μου γνώμη. Είχαμε μια πολύ καλή πρόταση. Πιστεύω πως οι νέες αυτές ρυθμίσεις θα μας πάνε μπροστά προς μια πολιτική κατευθυνόμενη, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα με καλύτερη διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φυσικά και ημών με ύψιλον. Οι στρατηγικές μας λοιπόν καλύπτουν όλα τα διευθυντικά ταμεία και υπάρχουν πολλές επιμέρους προτάσεις για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες που μας προσφέρονται. Αναφέρονται τα κίνητρα, αναφέρεται η αρεσιμότητα, πράγματα τα οποία πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά και να επικεντρώνονται σε ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Συγχρόνως όμως πρέπει να υπάρχει περιθώριο για προσαρμογές ανάλογα με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε, που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος και σας εύχομαι καρποφόρες συζητήσεις στη συνέχεια των ημερίδων αυτών. Και μην ξεχνάτε ότι του χρόνου στην ε, Επιτροπή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εισηγητές μας θα συνεχίσουν να δουλεύουν σε συνεργασία μαζί σας. Οπότε μην διστάσετε. Ό,τι θέλετε να συζητήσουμε μαζί, ελάτε να το συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο η Κομισιόν ανοιχτή σε εσά και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας θα Πριν κλείσουμε, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους. Είχαμε τεράστια ύλη να καλύψουμε, τα καταφέραμε. Σα ευχαριστώ όλου. Ευχαριστώ και του διερμηνεί, λέω Ξέρω ότι μερικέ φορέ όταν με βγαίνει ο χρόνο μιλάω όλο και πιο γρήγορα, οπότε ζητώ συγγνώμη. Η συζήτηση αυτή σίγουρα θα συνεχιστεί και του χρόνου. Είπατε ideas. Να, κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ πέρα ε, αυτές οι καρτούλες οι οποίες βοηθούν να κυκλοφορήσουν νέες ιδέες. Αν δείτε μια τέτοια καρτούλα, πάτε την, συμπληρώστε την με τις ιδέες σας. Ε, καλή συνέχεια.